Okay, good morning, dear colleagues. We um, Καλημέρα σα. Οι διερμηνεί σα πληροφορούν με τα λύπη ότι συνεχίζει η διεργασιακή διαμάχη με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι νέε συνθήκε εργασία, που αποτέλεσε το αντικείμενο προειδοποίηση για απεργιακή κινητοποίηση. Δυστυχώ λόγω τη εργασιακή διαμάχη η διερμηνία θα σταματήσει στι 12.30 ακριβώ όπω προβλέπει το πρόγραμμα τη συνεδρίαση. Περνάμε τώρα στην έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Εγκρίνεται και στι ανακοινώσει του Προέδρου. Έχουμε την απόφαση των συντονιστών στις 25 και 26 Απριλίου να υπάρξει η προθεσμία για τροπολογίε ε, για την πρόταση τη Κομισιόν για το θέμα του ΠΔΕΛΤΑΠ και δεν θα υπάρξει γνώμοδότηση. Προθεσμία των τροπολογιών θα ισχύσει για τα μέλη τη επιτροπή μας και μετά θα ψηφίσουμε. Οι σχετικέ ε, τροπολογίε θα αποτελέσουν την τελική γνωμοδότηση. Η συγητής θα είναι ο πρόεδρο και θα υποβληθεί στην Επιτροπή Αλίας ε, πριν ψηφιστεί εκεί. Οπότε η προθεσμία είναι 14 Ιουνίου 11 η ώρα. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας αναμένεται 9 και 10 Ιουλίου. Κατόπιν, προθεσμία τροπολογίας για την εφαρμογή την έγκριση της οδηγίας έγκρισης τύπου για δικυκλά και τρικυκλά και μοτοσυκλέτες στις 25 Απριλίου. Οι συντονιστές αποφάσισαν να δοθεί προθεσμία για τροπολογίες. Θα ισχύσει η ίδια διαδικασία όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Προθεσμία για τροπολογίες 19 Ιουνίου στις 11 η ώρα. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 13 Σεπτεμβρίου και στην ΙΜΚΟ στις 10 ε, και 11 Οκτωβρίου. Η τρίτη ανακοίνωση εργαστήριο για την ψηφιοποίηση και τα μαζικά δεδομένα για, από την ομάδα εργασίας για την υγεία την ηγεσία του Αλόης και της Σολεδάδ θα συνεδριάσει 19 Ιουνίου 10 έως 12 όλα τα μέλη της Επιτροπής μας ε, είναι προσκεκλημένα. Κατόπιν έχουμε ακύρωση τη απογευματινής συνεδρίασης 22 ε, και 23 Ιουνίου. Οι πρωινέ συνεδριάσεις παραμένουν και θα διανεμηθεί σύντομα η ημερήσια διάταξη. Καθιστώς στη διερμηνία. Στη διερμηνία έχουμε σε 20 γλώσσες. Ε, δεν υπάρχουν ε, εστονικά, λετονικά, μαλτέζικα και ιρλανδικά. Και όσον αφορά την διερμηνία έχουμε και μία ανακοίνωση από τους διερμηνείς. Οι διερμηνείς σας πληροφορούν τα λήψη τους ότι συνεχίζει η εργασιακή διαμάχη με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις νέες συνθήκες που αποτέλεσε το αντικείμενο προειδοποίηση για πυριακή κινητοποίηση. Η ποιότητα της διερμηνίας για ευρωβουλευτές και τους πολίτες κινδυνεύει. Δυστυχώ, Λόγω της διαμάχης αυτής, η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώς στις 12.30 ε, όπως προβλέπει το πρόγραμμα. τα περί μετάδοση στο διαδίκτυο ισχύουν ως συνήθως, όπως επίσης και τα της εφαρμογής ε, e-meeting. Κατόπιν έχουμε τις ανακοινώσεις της συνεδρίασης της 16ης Μαΐου. Τα έχετε λάβει ηλεκτρονικά, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις τότε εγκρίνονται έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 19 και 20 ε, Φεβρουαρίου. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος συνεδρίας εγκρίνονται. Μετά έχω κάποιες ε, ενημερώσεις ε, για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις για πέντε διαφορετικά ζητήματα. Πρώτα έχουμε κτηνιατρικά φάρμακα. Στις 15 ε, Μαΐου συναντηθήκαμε το Συμβούλιο και εστιάσαμε στην εναρμόνιση της σύνοψης των χαρακτηριστικών προϊόντων πέρα από τα ζητήματα του άρθρου 70 το ζήτημα 3 ομοιοπαθητικά φάρμακα αμοιβαία μέτρα για εισαγόμενα προϊόντα και αξιολόγηση περιβαλλοντικών αντικτύπων και επίσης ε, το θέμα του παραλλήλου εμπορίου και των ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση. Ο έκτος και τελευταίος ε, άτυπος ε, διάλογος έγινε στις 5 Ιουνίου. Εκεί πέρα Συμβούλιο Κοινοβουλίου και Κομισιόν κατέληξαν στις τελικές διατάξεις για όλα τα ζητήματα. Η προκατακτική συμφωνία θα υποβληθεί στην Κόρεπερ για έγκριση στις 30 Ιουνίου και θα ψηφιστεί στην Επιτροπή μας στις 20 Ιουνίου. Δεύτερον, η διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, ο τρίτος άτυπος διάλογος για την Ενεργειακή Ένωση έλαβε χώρα στις 23 Μαΐου. Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν συμφώνησαν σε πολλές διατάξεις που συζητήθηκαν σε τεχνικό επίπεδο και συζητήσαμε τέσσερα, τέσσερις δέσμες ζητημάτων σημειώθηκε σημαντική πρόοδος για την πρώτη δέσμη ζήτηματων, την εσωτερική αγορά ενέργειας και την ενεργειακή φτώχεια. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία στην ενεργειακή ασφάλεια και συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο για τα υπόλοιπα τρία ζητήματα και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επίσης συμφώνησαν σε μια εντολή για να μυστικοποιηθεί το κείμενο για την διαφάνεια στην χρηματοδότηση των μέτρων για το κλίμα και επίσης τα θεσμικά όργανα σημείωσαν πρόοδο στο ζήτημα της μακροπεριφερειακής συνεργασίας και οι περιτεροδιατάξεις παραπέμφθηκαν στο τεχνικό επίπεδο. Τρίτον, έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ο δεύτερος άτυπος ε, διάλογος για την έδρα της υπηρεσίας αυτής έλαβε χώρα στις 22 Μαΐου. Συμφωνήθηκε η ανάγκη να ολοκληρωθούν σύντομα διαπραγματεύσεις για να συνεχίσει η ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Καταλήξαμε στις ε, προσωρινές ε, τροπολογίες και έγινε μια παρουσίαση των Κομισιών σχεδίου προτάσεων για τις τροπολογίες 4 και 6. Το Κοινοβούλιο επανέλαβε το αίτημά του είναι μια πολιτική δέσμευση από όλα τα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στην αναθεώρηση της διαδικασίας επιλογής εδρών για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και να εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλες τις φάσεις κατά την άποψη του Κοινοβουλίου τα δύο εκτιμώντας ε, της ε, Προεδρίας για την διαδικασία δεν αποτελούν μια ικανοποιητική απάντηση στο αίτημα αυτό. Τέταρτον, ορισμός, ε, παρουσίαση και σήμανση των ίνοπνευματοδών ε, και γεωγραφικές ενδείξεις. Στον πρώτο άτυπο διάλογο στις 23 Μαΐου το Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν είχαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, για τις προτεραιότητες και τις κύριες πτυχές των θέσεων του Η συζήτηση ήταν επικοδομητική και ήδη στο θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων υπήρξε μια συνεννόηση για πιθανή ε, συμφωνία δεδομένων όμως των τεχνικών πτυχών και η Προεδρία και το Κοινοβούλιο αποφάσισαν να αναβάλουν στο τεχνικό επίπεδο την προετοιμασία του επόμενου διαλόγου που θα γίνει στις 27 Ιουνίου. Και τέλος, προώθηση των, ε, της ανανεώσιμης ενέργειας τέσσερις ε, κύκλοι συναντήσεων έγιναν. Ε, η Ήτρα είναι η επικεφαλής επιτροπή. Είχαμε μία παρουσίαση των αντίστοιχων εντολών. Ε, στην δεύτερη συνάντηση είχαμε ζητήματα αρμοδιότητας Ήτρε. Η ΕΝΒΗ έχει, ζητή, έχει αρμοδιότητα για ζητήματα αηφορίας και αερίων του θερμοκηπίου, το πλαφόν στις εκπομπές των μεταφορών, βιοκαύσιμα και διάφορους ορισμούς. Στον τρίτο τριμερή διάλογο 17 Μαΐου το Συμβούλιο έκανε συμβαστικές προτάσεις για την ιεραρχία των ρήπων και τα διαφορετικά κατόφλια που υπάρχουν στα κριτήρια φορής. Κατόπιν ο εισηγητής τόνισε την πολιτική σημασία των θέσεων του Κοινοβουλίου στους παραγράφους 8 και 10 και τις ε, πληροφορίες για την προέλευση των βιοκαυσίμων όλες οι αποφάσεις για τα άρθρα 26, 27 και 28 παραπέμφθηκαν στο τεχνικό επίπεδο. Η τέταρτη συνεδρίαση έγινε στις 6 Ιουνίου. Συμφωνήσαμε σε μια οριστική μορφή του άρθρου 27 και μια συζήτηση σε έναν πιθανό συμβασμό για εγκαταστάσεις συμπαραγωγής. Εξετάσαμε τις πιθανές διατάξεις βιοκαυσίμων μεταξύ άλλων και την επόμενη εβδομάδα στο Τρασβούργο θα έχουμε την επόμενη συνεδρίαση Αυτά λοιπόν από τις διαπραγματεύσεις και περνάμε στο επόμενο θέμα μια κοινή συζήτηση, παρουσίαση της συζήτησης της μελέτης, με συγχωρείτε, του Κέντρου Ερευνών του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της έκθεσης για τα προϊόντα φυτοπροστασίας ε, και του σχετικού κανονισμού. Η είναι ο κ. Πότς, ο αντιπρόεδρος μας. Όσον αφορά την ε, συζήτηση θα δώσω τον λόγο πρώτα απ' όλα στην υπηρεσία ερευνών ε, στην κυρία Καραμφίλοβα για 15 λεπτά και μετά θα συνεχίσει ο κύριος ε, Πότσο και μετά οι ομάδες και οι βουλευτές μπορούν να μιλήσουν. Uh, um, Εφόσον οι Άγκρη ΠΕΣΚ είναι επίσης υπεύθυνε επιτροπές για το θέμα, τα μέλη αυτής έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν, τα μέλη αυτών των επιτροπών μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Η PRS, η κυρία Καραφίλοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, είναι χαρά να σας παρουσιάζω εκ νέου το έργο της Επιτροπής Έρευνας του Τη Υπηρεσία Έρευνα του Κοινοβουλίου. Πέμπτη μελέτη που είμαστε η μονάδα μας για να στηρίξουμε την ΕΜΒΗ για τις διάφορες εκθέσεις ε, εφαρμογή. Βασιζόμαστε σε στοιχεία που υπάρχουν και παραγόμενα. Και γι' αυτό η μελέτη μας δίνει νέα στοιχεία. Ευχαριστώ όσου συμμετείχαν στη συλλογή στοιχείων. Επίση ευχαριστώ τους εξωτερικού ερευνητέ που επεξεργάστηκαν τα διάφορα θέματα. Βλέπετε τα ονόματά τους επί της οθόνης για λόγους χρονικούς δεν μπορούν να παρουσιάσουν το έργο τους. Οπότε θα προσπαθήσω τις 500 σελίδες της ενδελεχούς έρευνας να τις ε, παρουσιάσουν συντομία. Ποιο είναι το πρόβλημα το εφαρμοστικό με τον κανονισμό. Οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Να εξηγήσω ποιοι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί και για ποιο λόγο. Ο κανονισμός θέλει να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα τα φυτογενομικά προστασίας των φυτών είναι ασφαλή για το περιβάλλον και για την υγεία και πρέπει να λειτουργεί και εύρυθμα εσωτερική αγορά με αυτά τα προϊόντα και να βελτιωθεί και η γεωργική παραγωγή. Θεωρήσαμε ότι αυτοί οι στόχοι δεν καλύπτονται. Ποιο ο λόγος. Είναι το πώς τα μέσα του κανονισμού χρησιμοποιούνται. Και αυτά τα μέσα είναι πρώτα απ' όλα η έγκριση των ουσιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεω, Δεύτερον, η εθνική αδειοδότηση των προϊόντων και προστασία των φυτών χρησιμοποιώντα τι συγκεκριμένε ουσίες. Και τρίτον, η επιβολή του νόμου σε εθνικό επίπεδο. Θα ξεκινήσω από τις ε, διαδικασίες εγκρίσεως. Να εξηγήσω και τις διάφορες φάσεις, διότι αυτό θα βοηθήσει την κατανόηση των πορισμάτων διαδικασία. Ξεκινάμε την αξιολόγηση τη ουσία, για τυχόν κινδύνου ε, σύμφωνα με τα κριτήρια του κανονισμού. Είναι τα ε, κριτήρια αποκοπής. Αν δεν δείξουν κίνδυνο, ότι δημιουργούν κίνδυνο οι ουσίες, αξιολογούνται για το κίνδυνο που μπορεί να προξενήσουν. Οι κίνδυνοι λοιπόν αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης μπαίνουν σε μια έκθεση αξιολογήσεως που εξετάζεται από μοτίμους από την Υπηρεσία Ασφαλείας Τροφίμων. Και μετά αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί των ε, διαφόρων κινδύνων. Μετά από περίπλοκη διαδικασία λαμβάνεται η απόφαση. Συμμετέχουν εμπειρογνώμονε από κράτη-μέλη που συμμετέχουν στη μόνιμη επιτροπή των φυτών, ζωοτροφών. Είναι η Επιτροπή Επιτροπολογίας ΠΑΦ. Να δούμε τώρα λοιπόν ποιες, ε, πώς γίνεται η έγκριση των ουσιών. Πρώτα απ' όλα γίνεται επιστημονική αξιολόγηση των ουσιών. Δεύτερον, η επίδοση των διαφόρων αρμοδίων εθνικών αρχών. Και τρίτον, εξετάζεται η διαφάνεια της διαδικασίας. Όσον αφορά την επιστημονική εξολόγηση των ουσιών, υπάρχει ένα θέμα με την εναρμόνιση. Η εναρμόνιση έχει βελτιωθεί σε κάποιους τομείς, όπως είναι η τοξικολογία, όμως είναι ατελής σε άλλους τομείς, όπως η οικολογική τοξικολογία. Οι εξολογητές δεν μπόρεσαν να αξιολογήσουν πλήρως τις ουσίες και τι κινδύνους δημιουργούν, κάτι που απαιτεί ο κανονισμός. Ποια είναι τα αποτελέσματα. Αρνητικές συνέπειες για την υγεία, το περιβάλλον και την προστασία της γεωργίας. Άλλο πρόβλημα με την εναρμόνιση. Κάποια κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν τους προσανατολισμού που δεν είναι νομικά δεσμευτικοί. Έτσι δημιουργείται κάποια βεβαιότητα για τους ετούντες. Δεν ξέρουν με τι να συμμορφωθούν. Τα αποτελέσματα αξιολογήσεως εξαρτώνται από την αρμόδια αρχή που εξετέλεσε την αξιολόγηση. Αυτό δεν έπρεπε να γίνεται διότι εδώ αντιβαίνουμε το σκοπό της εναρμονήσεως. Θέλουμε να εφαρμόζονται παντού οι ίδιες προδιαγραφές όλα τα κράτη-μέλη. Άλλο πρόβλημα για την εξολόγηση των ουσιών. Η εξολόγηση των προϊόντων, πώς εφαρμόζεται την πράξη. Τι προβλήματα διαβλέπουμε. Πρώτο, προσέγγιση βάση κινδύνου δεν υποστηρίζεται από αυτούς που εξετάζουν το ρίσκο, ακολουθούν το ρίσκο. Η αξιολόγηση της γλυφοσάτης. Δεν ξέρουμε αν η αξιολόγηση έγινε σωστά και από ανεξάρτητο φορέα. Τρίτον, η γλυφωσάτη δημιουργεί το ερώτημα. Ποιος παράγει τα προς στοιχεία. Οι αξιολογήσεις τώρα γίνονται ε, βάσει αποκλειστικά ε, στοιχείων που δίνουν οι ετούντες. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες, λόγω χρόνου. Κοιτάξτε τα πορίσματά μας που είναι στην ε, μελέτη. Δεύτερη πτυχή της διαδικασίας εγκρίσεως. Η επίδοση των εθνικών αρμοδίων αρχών. Οι περισσότερες, όχι όλες οι αρμόδιες αρχές, έχουν τη δυνατότητα να είναι εισηγητές των κρατών μελών και να δώσουν αξιολογήσεις, εκθέσεις αξιολογήσεις στην ΕΦΣΑ. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ εθνικών αρμοδίων αρχών όσον αφορά τεχνογνωσία και προσωπικό. Όλες οι αρχές έχουν σοβαρό πρόβλημα ελλείψης προσωπικού και δεν γίνεται σωστά η κατανομή του φόρτου εργασίας αξιολόγησης. Αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των ουσιών. Και αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις στην όλη έγκριση. Και μετά σε εθνικές αδειοδοτήσεις ε, των προϊόντων που εμπεριέχουν τις συγκεκριμένες ουσίες. Η τεχνογνωσία και η διαφορετική στελέχωση των διαφόρων αρμοδίων αρχών οδηγεί σε διαφορά της ποιότητας των εκθέσεων αξιολόγησης. Έτσι περαιτέρω. Τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν συμμετέχουν στην έκθεση, την εξέταση των εκθέσεων από πλευρά ομοτήμων. Αυτή η διαδικασία εξετάσεως από ομοτήμους καλύπτει προβλήματα ποιότητας των εκθέσεων. Και αυτό εξαρτάται από τη συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία. Οπότε η ΕΦΣΑ δεν μπορούσε να κάνει σωστά τον έλεγχο ποιότητας. Προβλήματα είναι όλα αυτά. Όσον αφορά τι αρχές. Οπότε ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού φαίνεται ότι είναι κάτι αδύνατον. Αυτό έχει επιπτώσει για την υγεία και το περιβάλλον. Τρίτο σημαντικό θέμα, η διαφάνεια όσον αφορά το μέσο έγκρισης. Η διαφάνεια είναι προβληματική. στη φάση δραστηριότητας των αρμοδίων αρχών είναι προβληματική. Οι πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση ε, διατίθενται μόνο σε επίπεδο εξετάσεως ομοτήμων στο επίπεδο ΕΦΣΑ, όχι όμως πάντα φιλικά προς το χρήστη. Λείπει λοιπόν η διαφάνεια από όλα τα στάδια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότερες φορές η λογική πίσω από τις αποφάσεις για τη χείριση του κινδύνου και την ενημέρωση εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις ε, δεν δημοσιοποιούνται ανοιχτά Οπότε οι αποφάσεις καμιά φορά διαφέρουν από τις επιστημονικές συμβουλές που δίνονται από την ΕΦΣΑ και στους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Αυτό οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες για την υγεία και το περιβάλλον και το κοινό χάνει την εμπιστοσύνη του στο ρυθμιστικό σύστημα. Και η επικοινωνία ήταν προβληματική όσον αφορά τους κινδύνους. Πάω στο δεύτερο βασικό μέσο του κανονισμού. Η εθνική αδειοδότηση προϊόντων που εμπεριέχουν εγκεκριμένε ουσίες. Εξολόγηση των προϊόντων και αποφάσει περί κινδύνων λαμβάνονται αποκλειστικά σε επίπεδο κρατών μελών. Τα βασικά προβλήματα εφαρμογής σχετίζονται με την επιστημονική αξιολόγηση των προϊόντων. Κυρίω για την αξιολόγηση σωρευτικών αποτελεσμάτων, η επίδοση των αρμοδιών αρχών είναι προβληματική και η διαφάνεια. Θα εστιαστώ στι επιδόσει των εθνικών αρμοδίων αρχών και για τα θέματα διαφάνειας θα μιλήσω. Τι βρήκαμε. Ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης καθυστερεί όσον αφορά την αξιολόγηση και την ανάλυση των κινδύνων και δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες νόμιμες ε, προθεσμίε. Υπάρχουν βασικοί λόγοι για τις καθυστερήσεις. Πρώτα απ' όλα, οι αρχές δεν έχουν αρκετούς πόρους. Δεύτερον, ο φόρτος εργασίας της αξιολογήσης δεν μοιράζεται ε, δίκαια ανάμεσα στις αρχές και οι αρχές δεν εμπιστεύονται τις αξιολογήσεις ημέν των δε όσον αφορά τα προϊόντα. Όλα αυτά δημιουργούν στρέβλωση εσωτερικής αγοράς και πρόβλημα με την αμοιβαία αναγνώριση των αξιολογήσεων. Η καθυστέρηση αδειοδότησης δημιουργεί προβλήματα. Και καμιά φορά ε, εγκρίνονται από τα κράτη-μέλη προϊόντα περιέχουν ουσίες που έχουν αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Το άρθρο 53 του κανονισμού οδηγεί σε κατεπίγουσες αδειοδοτήσει δυνάμει του άρθρου 53, γιατί αν έχουν καθυστερήσει οι αξιολογήσεις. Τι είδαμε, ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το άρθρο 53 χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη αντίθετα με τις προθέσεις του νομοθέτη. Τις λεπτομέρειες στην έκθεσή μας. οι πτυχές διαφάνειας της αδειοδότησης προϊόντων υπάρχουν. Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών και η πρόσβαση στα στοιχεία για τη διαδικασία και τα στοιχεία είναι περιορισμένη. Οπότε το ευρύτερο κοινό δεν κατανοεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Τέλος η επιβολή, η υλοποίηση του κανονισμού ε, και το σχετικό μέσο του κανονισμού, το τρίτο. Τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αγορά και η χρήση τους από τους χρήστες δεν συμμορφώνται απαραίτητα με τους όρους αδειοδότησης όσον αφορά σύνθεση και χρήση. Αυτό ισχύει για προϊόντα που παράγονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εισάγονται και από τρίτε χώρε. Τα προβλήματα συμμόρφωση οφείλονται σε επιδόσει των εθνικών αρχών αλλά και σε κενά του κανονισμού. Προβληματικοί έλεγχοι σε εθνικό επίπεδο υπονομεύουν σημαντικά την επίτευξη των τεσσάρων στόχων του κανονισμού. Και αυτό έχει αρνητικέ συνέπειε στην υγεία, το περιβάλλον, την αγορά και την προστασία των γεωργικών προϊόντων και τη γεωργία γενικότερα. Εν κατακλείδη, όπω βλέπετε, η υλοποίηση και η χρήση του κάθε ενό από τα τρία μέσα είναι προβληματική και τα προβλήματα ξεπερνούν την αξιολόγηση συγκεκριμένων ουσιών. Και εδώ έρχεται το μήνυμά μου σήμερα το πρωί για σας. Είναι μεγάλη μόνο η γενική εικόνα της εφαρμογής και υλοποίησης θα μπορούσε να είναι κάτι χρήσιμο για να ενημερώσει τις συζητήσεις. Η εξολόγηση που έκανε το EPRS σας δίνει αυτή την εικόνα την περιπλοκή. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία της δουλειάς μας. Έχουμε κάνει συστάσεις για δράση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και καλείστε να δείτε τις συστάσεις στη μελέτη μας. Κλείνω εδώ. Ευχαριστώ την προσοχή σας. Μαζί με την ερευνητική ομάδα μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Η Δ. Λίβια Χάμπλιν και η κυρία Εύελιν Underwood δεν μπορούσαν να έρθουν, ζητούν συγγνώμη, αλλά είναι διαθέσιμες. Μπορούν να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις. Γραπτός. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Πότσο, ο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλημέρα, συνάδελφε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Εκατερίνα όχι μόνο για την εξαιρετική παρουσίασή της, καθώς ε, κατάφερε να παρουσιάσει συνοπτικά το έργο έξι μηνών σε 5-10 λεπτά, αλλά να την ευχαριστήσω επίσης για την προσωπική της συμβουλή στη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Επίσης ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο της ομάδας των υπηρεσιών ε, μελέτησης ε, του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτήν την έκθεση αξιολόγησης εφαρμογή του κανονισμού που υπερβαίνει τις 500 σελίδες. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι αργότερα σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε κάποια ερωτήματα ε, και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να το κάνετε. Συχνά αναφερόμαστε στην ανάγκη του να ακολουθούμε ε, τα ε, τελευταία επιστημονικά πρότυπα και ήρθε η ώρα να το αποδείξουμε. Και θα πρέπει λοιπόν ε, να λάβουμε υπόψη μας τα όσα έχουν προβλεφθεί σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες και τις προθεσμίες και στο πλαίσιο της δικής μας αλλά και στο πλαίσιο της Επιτροπής ε, ΠΕΣ. Και ουσιαστικά μια αξιολόγηση σε ό,τι αφορά αυτόν τον ε, κανονισμό γίνεται για πρώτη φορά, πράγμα το οποίο είναι κάκιστο. Το ότι δηλαδή μετά από 10 χρόνια για πρώτη φορά αξιολογούμε τον τρόπο εφαρμογής αυτού του κανονισμού. και ε, καθώς η Επιτροπή προβαίνει αυτή την περίοδο ε, σε μια αναθεώρηση της γενικής νομοθεσίας στο πλαίσιο του σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα, η διαδικασία που ακολουθεί είναι πιο περιορισμένη, ενώ εδώ ακολουθούμε τα, και εφαρμόζουμε τα τελευταία επιστημονικά πρότυπα. Επίσης, εδώ έχω λάβει υπόψη μου και όλα τα σχετικά πορίσματα άλλων μελετών και αποφάσεων του δικαστηρίου. Κατά τη σύνταξη της ε, έκθεσής μου, περιορίστηκα ε, φυσικά σε ό,τι αφορά και τη σχετική δήλωση αλλά και την ε, ε, έκθεση στα σχετικά όρια, οπότε περιορίστηκα στα σημεία που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, της ΕΝΒΕ. Ε, καθώς δεν μπόρεσα να καλύψω τα πάντα, θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες, αλλά θα ήθελα βέβαια να μείνει σύντομη και περιεκτική αυτή η έκθεση. δεν μπορούμε δηλαδή σε μια τέτοια έκθεση να περιλάβουμε τα πάντα έτσι ώστε ουσιαστικά να περιλαμβάνει σωρία στοιχείων χωρίς να δίνει ένα κύριο μένωμα. Ε, οι επιτυχίες ε, που αφορούν την ε, Επιτροπή Άγκρη θα αναλυφθούν από εκείνη και θα ψηφίσει τότε στι 20 Ιουνίου για αυτά τα ζητήματα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που εγώ θίγω, υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού, καθώ ο κανονισμό προβλέπει στενή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν επί χάρτου ένα πολύ καλό κανονισμό αλλά οι στόχοι του οποίου έχουμε θέσει σε ό,τι αφορά και την υγεία και το περιβάλλον δεν επιτυγχάνονται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, τόσο ώστε να εφαρμοστεί σωστά ο κανονισμό. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ιδιαίτερα ότι ε, ανεπαρκής ε, εναρμόνιση των δεδομένων σε ορισμένου επιστημονικού τομεί μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικέ συνέπειε για την υγεία και το περιβάλλον. Από εκεί και μετά υπάρχει πρόβλημα σε επίπεδο διαφάνεια. Διαφάνεια σε ό,τι αφορά ε, τι ε, διάφορε φάσει τη διαδικασία έγκριση. Κάτι το οποίο και αυτό με τη σειρά του έχει ανητικές συνέπειες για, την υγεία ε, και το περιβάλλον, αλλά δημιουργεί και δυσπιστία του εκείνου σε ό,τι αφορά ε, την, ε, το δικό μας σύστημα για την έγκριση των φυτοφαρμάκων. Και γι' αυτό χαιρετίζω και την πρόταση και τη σχετική έκθεση σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα της χρήσης των φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, ορισμένα κανονιστικού χαρακτήρα ζητήματα δεν καλύπτονται από τη σχετική πρόταση ειδικότερα σε ό,τι αφορά την διαδικασία αξιολόγηση του κινδύνου την οποία διεξάγει η ΠΑΦ. Ε, και η διαδικασία τη έγκριση των σχετικών δραστικών ουσιών θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Ε, τρίτον, θα πρέπει να περιορίσουμε τι ε, εξαιρέσει, τι παρεκκλήσει που παρέχονται στα κράτη-μέλη υπό το άρθρο 53. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γίνεται κατάχρηση αυτή τη εξαίρεση, ώστε τα κράτη-μέλη να καταστατηγούν ουσιαστικά την νομοθεσία. Η αξιολόγηση καταδεικνύει ότι το άρθρο 53 εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη ε, με διαφορετικό τρόπο ε, ε, διαφορετικό από αυτό που προέβλεψε ο νομοθέτης. Ουσιαστικά δηλαδή το 2016 και μόνο 123 εξαιρέσεις δόθηκαν. Ενώ έχουμε και την ε, μερική, το παράδειγμα της μερική απαγόρευσης των νέων νοικοτινοειδών ακριβώς επειδή πολλά κράτη-μέλη αξιοποίησαν το άρθρο 53. Από εκεί και μετά υπάρχουν μία σειρά από περαιτέρω ζητήματα πέραν αυτών των βασικών προτεραιοτήτων και τα αναφέρω επί τροχάδι. Η ανάγκη τη χρήση ε, ε, καλών αγρονομικών πρακτικών και, και η χρήση εναλλακτικών προϊόντων, η ανάγκη εφαρμογής αξιολόγησεων επιβεβαίωσης η ε, ανάγκη ε, επιβολής ε, κοινών ελέγχων αλλά και η ανάγκη ελέγχου των μειγμάτων διαφορετικών φυτοφαρμάκων. Παρά τα, τις, τα, τα ελλείμματά της, αυτός ο κανονισμός αποτελεί την καλύτερη νομοθεσία που έχουμε σε αυτό το τομέα και συμφωνώ πλήρως με το συμπέρασμα ότι η δράση που θα πρέπει να αναλυθεί στον τομέα της φυτοπροστασίας θα πρέπει να αναλυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο κανονισμός πραγματικά επιτυγχάνει τους στόχους του σε ό,τι αφορά την υγεία ε, και το περιβάλλον και ότι λαμβάνει υπόψη την αρχή της ε, προφύλαξης ε, και καλύπτει κυρίως και προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως οι έγκυες, οι γυναίκες, τα βρέφη και τα παιδιά. Τώρα επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να αναφερθώ στο χρονοδιάγραμμα. Παρά την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων να υπάρξει μια αναβολή της σχετικής προθεσμίας μετά από τη διαβούλευση που έκανα διμερός και με τους εστιώδεις να επιμείνω στο αρχικό χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή να γίνει ψηφοφορία εδώ στην ένβηση στις 10 Ιουλίου. Και αυτό γιατί η απόφαση τελικά για αναβολή τη ε, προθεσμία από διάσκεψη των προέρχων ε, ήρθε ε, καθυστερημένα και κατά συνέπεια δεν είχαμε και την κατάλληλη προθεσμία σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση τη μετάφραση. Οπότε δεν υπάρχει τη σήμερον ημέρα, λόγω και του χαμηλού αριθμού τροπολογιών, να παραταθεί η διαδικασία. Καλό είναι βέβαια ταυτόχρονα να οριστικοποιήσουμε, να εγκρίνουμε αυτή την έκθεση από την πλευρά της ΕΝΒΗ πριν από το θερινό διάλειμμα. Αυτά από την πλευρά μου και σας ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε τη δυνατότητα να κάνω αυτή την παρουσίαση και αναμένω με ενδιαφέρον τα σχόλια που θα κάνουν τόσο οι συνάδελφοι όσο και οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ τον ε, εισηγητή. Περνάμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Κάποιοι ακόμα δεν έχουν προσέλθει. Βλέπω πως ο κύριος Χόισλινγκ είναι ο πρώτος από τους συζητητές που έχουμε εδώ μαζί μας. Ε, θα του δώσω τώρα το λόγο. Και αν ε, καταφτάσουν και σκιώδες συζητητές από τις ε, υπόλοιπε πολιτικές ομάδες, θα τους δώσω φυσικά τις αυτούς το λόγο. Ο κύριος Χόισλινγκ έχει το λόγο. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση. Είναι νομίζω θετικό το ότι έχουμε καλή νομοθεσία αλλά δεν εφαρμόζεται επαρκώ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το έλλειμμα δράσης σε πολλούς ε, τομείς και βεβαίως εδώ πέρα ως συνήθως ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αναφέρατε το θέμα της γλυφοσάτης, εκεί πέρα είναι σαφές ε, ποιες είναι οι ελλείψεις στο σύστημα και πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό χαιρετίζουμε και εμείς ξεκάθαρα την πρωτοβουλία διαφάνειας της Κομισιόν. Τώρα, εάν πηγαίνει αρκετά μακριά, είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί από εκείνο. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούσε να πηγαίνει ακόμα παραπέρα. Ειδικά το θέμα της διαφάνειας είναι πολύ ευαίσθητο. Αλλά πρέπει τελικά να δούμε το ερώτημα του τι γίνεται με το υφιστάμενο δίκαιο σε περιπτώσεις εξαιρέσεων όπως ε, προβλέπει η παραγραφός 50 αναφέρθηκε το ζήτημα των ε, νεονικοτινοειδών ε, που δεν μας είχε απασχολήσει γιατί είχαν ζητήσει εξαιρέσεις οι οποίες ελάμβαναν χωρίς κανένα πρόβλημα. δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή όταν απαγορεύουμε μια ουσία εγώ αναμένω να πέφτει η χρήση της και πολύ συχνά μετά δίνουμε πάρα πολύ εύκολα εξαιρέσει. Πρέπει λοιπόν να αντιδρούμε τότε και δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το γεγονό ότι έχουμε λίγους ειδικού είναι γνωστό αυτό και στην ΕΦΣΑ και τίθεται βεβαίως και το ζήτημα της ανεξαρτησίας των ειδικών που πρέπει να συζητηθεί. Και πέρα λοιπόν χρειαζόμαστε περισσότερους ειδικού, ε, ανεξάρτητους ειδικού στα κράτη-μέλη, στα διάφορα πάνελ ε, της ΕΦΣΑ για να έχουμε λογικές διαδικασίες και βεβαίως ε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε 27 χώρες να εφαρμόσουν τελικά τον κανονισμό διαφορετικά. Πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση αναφέρθηκε. Νομίζω και συμφωνώ πλήρως με αυτό ότι ένα εξετάμενο κανονισμό πρέπει να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την ελλειπή εφαρμογή και τελικά να έχουμε κινδύνους για το περιβάλλον και τον καταναλωτή. Γι' αυτό κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει συζήτηση περί αλλαγής ε, του νόμου και να δούμε και στην Επιτροπή ΠΕΣ ε, πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ε, θα έλεγα να υπάρξει μια εναρμόνιση και μετά να δούμε τα επόμενα κοινοβουλευτικά βήματα. Αλλά συμφωνώ με τον συναδελφό και να ψηφίσουμε κατόπιν γρήγορα στις 12 ε, του μηνός. Έχουμε λίγο χρόνο και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος ε, Πελτσίνη. Ευχαριστώ. Εγώ συναρμολογώ τα κομμάτια από αυτά που άκουσα. Να υπενθυμίσω, χρειάστηκαν πέντε χρόνια διαβουλεύσεων πριν να έχουμε μια πρώτη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατέφθασε μόλις το 2006 και μετά χρειαστήκαμε άλλα τρία χρόνια για να τεθεί σε ισχύ και από το 2009 μέχρι σήμερα πέρασαν άλλα δέκα χρόνια. Ίσως και γι' αυτό πέρσι ένα εκατομμύριο πολίτες υπέγραψαν μία πρωτοβουλία πολιτών για να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο που τη γλυφοσάτη, αλλά να μεταρρυθμίσει όλη τη διαδικασία διοδότησης των παρασιτοκτόνων. Το θέμα των παρασιτοκτόνων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ την κοινή γνώμη. Οι πολίτες έχασαν την εμπιστοσύνη απέναντι στους θεσμούς και στους επιστημονικούς οργανισμούς που θα έπρεπε να δώσουν απαντήσεις. Για, την για τον εντοπισμό των κινδύνων που αφορούν μια... τη χρήση μιας συγκεκριμένης ενεργού ουσία. Ακούσαμε ότι χρειάζεται βελτίωση και διαφάνεια. Αλλά όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές εθνικού επίπεδο, αυτά που συμβαίνουν εκεί παραμένουν μυστήριο. Δεν ξέρουμε πόσα αιτήματα για διοδότηση έχουν υποβληθεί και ποια φυτογειονομικά ε, προϊόντα έχουν αδειοδοτηθεί. Δεν ξέρουν οι πολίτες εάν τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν συχνά παρεκκλήσεις, δεν έχουν ιδέα από αυτού. Παρεκκλήσεις που επιτρέπει η νομοθεσία για κατεπίγουσες ανάγκες. Αλλά μέσω στρέβλωσης διατίθενται προϊόντα στην αγορά που έχουν αποδεδειγμένα επιζήμια συνέπεια επιρροή στην υγεία και στο περιβάλλον. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έχει εργαλεία για να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας, ως εγγυητής όσον αφορά αυτά τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκοντίν, επόμενο και ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση του, του κ. Πόκ όσον αφορά το κανονισμό για, για τα προϊόντα τα φαρμακο-υγειονομικά δείχνουν πως η αξιολόγηση είναι δυσλειτουργική καθώς και αδειοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυσλειτουργίες που σωρεύτηκαν όσον αφορά και το είδαμε στην αδειοδότηση της γλυφοσάτης. Ε, είναι πλήρως η διαδικασία. Και η Γερμανία βρίσκεται στη θέση ε, ε, κατηγορούμενο όσον αφορά τις δραστηριότητες της Bayer και της Monsanto και δημιουργήθηκε η Ειδική Επιτροπή για τα Παρασιτοκτόνα που ακόμα λειτουργεί για να εντοπιστεί η πηγή των προβλημάτων. Ο εισηγητή μα εξηγεί ότι η εφαρμογή του κανονισμού ε, δεν είναι αποτελεσματική και υπάρχουν δυσκολίε λόγω ελλείψεω διαφανεία και εναρμόνιση. και χρειάζεται περισσότερη εξουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καλύψει διαφορέ μεταξύ κρατών μελών. Στην πραγματικότητα τα αντιμετωπιζόμενα προβλήματα είναι πολιτικής φύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει αποφάσεις, δίνει τις, ε, ε, τις αξιολογήσεις στην ΕΦΣΑ για λόγους ιδεολογία. και όχι επαρκή αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη. Όπως και για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, βλέπουμε ότι χρειάζεται αλλαγή προσέγγιση όσον αφορά την επικινδυνότητα των παρασιτοκτόνων. Περίοδο που χρησιμοποιείται η ουσία ενώ ε, τελικά η έψα βασίζεται στη δόση και όχι στην χρονική διάρκεια χρήσεω ενό προϊόντος. Χρειάζεται τοξικολογία του 21ου αιώνα, ενώ η ΕΦΣΑ χρησιμοποιεί διαδικασίε τη δεκαετία του 60. Άρα υπόκειται σε πιέσει των διαφόρων βιομηχανιών και των λόμπι. Διαφωνώ με του συναδέλφου που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επαρκέ επίπεδο για την ε, δράση τη ρυθμιστική. Διότι στην πράξη η Ένωση απέδειξε ότι δεν ανταποκρίνεται στο ύψο των περιστάσεων. Αντίθετα, μια δράση σε ευρωπαϊκή κλίμακα είναι κάτι που απαιτείται μέσω ενό μοντέλου συνεργασία κρατών μελών. Να δίδεται το ίδιο βάρο σε όλου όσον αφορά την αξιολόγηση. Τα φυτογενομικά προϊόντα λοιπόν ε, που είναι ενδοκρινικοί διαταράχτες δεν αναφέρονται στην έκθεση. Δεν υπάρχουν επαρκείς ε, ε, ορισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σωστές διαδικασίες στην απαγόρευση των προϊόντων. Όσον φάει τις παρεκκλήσεις, που είναι πολλές και μας ανησυχούν, συμφωνώ με τους συναδέλφους. Πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των παρεκκλήσεων και δυνατότητα χρήσεως των παρεκκλήσεων. Διότι έτσι δημιουργείται στρέβλωση στην αγορά και μεταξύ κρατών μελών. Θα υποβάλλω τροπολογίε. Σύμφωνα τι οποίε τα κράτη-μέλη και οι εθνικοί φορεί θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο τη αξιολόγηση. Και θέλω να πω ότι σήμερα η νέα αγορά εμποδίζει τα κράτη-μέλη που θέλουν να απαγορεύσουν την επικράτειά του προϊόντα και ουσίε να ελέγξουν και απαγορεύσουν τα τρόφιμα που ήρθαν σε επαφή ή που συνδέονται με αυτά τα προϊόντα. Είναι κάτι που ε, δεν επιτρέπει την απαγόρευση. Ε, και επίσης υπονομεύει καμιά φορά και την ανταγωνιστικότητα κάποιων κρατών μελών, το υφιστάμενο πλαίσιο. Ευχαριστώ. Μου είπαν ότι εκ μέρου της Άλντε η κυρία Μιούλερ θα μιλήσει. Η... Και Φίτεμαρ μετά. Στην κυρία Μίλλερ δίνω πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, στο σχέδιο έκθεσή σας ε, λέτε πως ε, δεν είναι πάρα πολύ καλή αυτή η πρόταση, κάτι το οποίο μου προξενεί έκπληξη γιατί μας έχει απασχολήσει εδώ και καιρό και έχω συζητήσει πολλές ώρες με ειδικού ε, και ένας από τους πιο επικριτικούς από αυτούς λέει πως έχουμε το καλύτερο σύστημα αδειοδότησης στην Ευρώπη Νομίζω ότι θα πρέπει να το αναγνωρίζουμε ακόμα και αν δεν είναι όλα τέλεια. Και έχουν δίκιο οι προλαλήσαντες. Εδώ πέρα μιλάω ιδιαίτερως για τα μέσα φυτοπροστασίας στις τρεις ζώνες ε, και το σύστημα διοδότησης. Είναι καλή η νομοθεσία αλλά δεν λειτουργεί στο εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχει εναρμόνιση. Και βεβαίω ω σκιώδη εισηγήτρια στην Επιτροπή Γεωργίας Ήμασταν υπέρ βεβαίως μιας ρεαλιστικής αξιολόγησης ε, των θετικών και των αρνητικών και το ίδιο νομίζω θα κάνουμε και εδώ και σημαντικό για εμάς ε, στην Άλντε είναι να γνωρίζουμε ότι ε, πρέπει να υπάρχει ένας αποδεκτός κίνδυνος τον οποίο να αναγνωρίζουμε. Ναι, δεν αμφισβητούμε κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να υπάρξει και μία ανάλυση κόστους ωφέλους και να δώσουμε ιδιαίτερη βάση και προσοχή σε αυτό. Και βεβαίως υπάρχουν και πολλές ομάδες ουσιών που χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ ειδικέ περιπτώσεις. Φοβούμαστε δηλαδή ότι θα χαθούν αυτοί οι πολύ μικροί τομείς και αυτό το οποίο μας ενοχλεί είναι τα προϊόντα χαμηλού ρίσκου δεν ε, τα είχαμε εμείς ε, κατά νου, αλλά παρόλα αυτά θα περιληφθούν. Γενικά όμως θεωρούμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Έχουμε πολλές αλληλεπικαλύψεις με την Επιτροπή ΠΕΣΤ και ότι έχουμε πολλούς ειδικού ε, εκεί και πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή και πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ ήρθε και την, ήρθε η ομιλήτρια του ΕΛΚ που αντικαθιστά την κυρία Μαγκίνης, η κυρία Ντελάη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Μαγκίνη ζητεί συγγνώμη, διότι είναι στην ε, μέρα μελέτης ε, του ΕΛΚ. Θέλω να σας πω τα εξή. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα παρασιτοκτόνα είναι από τις πιο αυστηρές στον κόσμο. Αυτό υπόθηκε και από άλλο συνάδελφο. Ο κανονισμό που αφορά τα φυτογενομικά προϊόντα προφανώ το τμήμα αυτού. Συμπληρώνεται από την οδηγία για την χρήση τη βιώσιμη των παρασιτοκτόνων, τον κανονισμό για τα Βιοκτόνα κανονισμός για την νομοθεσία για τα τρόφιμα εν γέννη, την νομοθεσία για τα κατάληπτα των παρσιτοκτώνων και τον κανονισμό για τα χημικά προϊόντα. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτά τα θέματα είναι κάτι υποφελέ για όλου του μετέχοντε, είτε είναι οι πολίτε, τα κράτη-μέλη, αλλά και η βιομηχανία. Και είναι πραγματικά μια προστιθέμενη αξία να υπάρχει μια πολιτική παρασιτοκτόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ο κανονισμό για τα φυτογενομικά προϊόντα αποτελεί καθαρή βελτίωση σε σχέση με την πρώτερη νομοθεσία. Α, συγγνώμη. Ναι, να πάω πιο σιγά για τους διερμηνείς. Συζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, έλεγα ότι ο κανονισμός για τα φυτογειονομικά προϊόντα αποτελεί καθαρή βελτίωση σχετικά με την πρώτερη νομοθεσία. Παραδείγματο χάρη τα κριτήρια της αναστολής ε, ε, έχει εισαχθεί. Λοιπόν, οι ουσίες που είναι ε, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή ενδοκρινικοί διαταράκτες μπορούν να απαγορευτούν. Αυτό δεν ε, προβλεπόταν στην προηγούμενη νομοθεσία. Όμως, το, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος του κανονισμού. Τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν το σύστημα των ζωνών για την αδειοδότηση νέων προϊόντων. Επιπλέον, χρειάστηκε χρόνο ούτω ώστε ο ορισμό του όρου ενδοκρινική διαταράκτε να εξευρεθεί και αυτό ο ορισμό θα τεθεί σε ισχύ μόλι τον επόμενο Νοέμβριο για τα φυτογενομικά προϊόντα. Η νομοθεσία που απαγορεύει αυτέ τι ουσίε στα προϊόντα τα φυτογενομικά χρονολογείται όμω από το 2009. Άρα υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωση για την εφαρμογή του κανονισμού. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές από χώρα σε χώρα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές συμμορφώνονται με αυτόν τον κανονισμό ή όχι. Κάποια κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν παρεκκλήσεις από το άρθρο 53 περισσότερο από άλλα κράτη-μέλη. Ιδού λοιπόν τα βασικά διακυβεύματα του κανονισμού. Ε, είναι τρία αυτά, η ανεξαρτησία, η διαφάνεια, η έρευνα και η καινοτομία. Όσον αφορά την ανεξαρτησία, οι αρχές αξιολόγησης, εθνικές και ευρωπαϊκής, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και από τη βιομηχανία και από τους πολιτικούς. Χρειαζόμαστε πιο προθυμένη συζήτηση για το ποιος πληρώνει τις επιστημονικές μελέτες. Οι προτάσεις αλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την νομοθεσία για τα τρόφιμα που δίνουν τη δυνατότητα διοδότησης στην ΕΦΣΑ ε, χρειάζεται μελέτη, αλλά είναι πρόσδεκτη. Όσον αφορά τη διαφάνεια, η διαφάνεια είναι ουσιαστική για να εξασφαλίζεται και να ενθαρρύνεται η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Πώς να εξασφαλιστεί η διαφάνεια χωρίς να επιφορτιστούν, ε, να βάλουμε πολύ άχθος στους επιστήμονες, είναι κάτι που εξεταστεί. Οι αρμόδιες αρχές, οι εθνικές, χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη για τη σύνταξη εκθέσεων, ούτως ώστε να είναι πιο ευανάγνωστος. Τέλος, εάν κάποιες αυτές τις εκθέσεις γίνουν προσβάσιμες επιτρέπει να, διασκεδάσουν, να διασκεδαστούν οι ανησυχίες του κοινού. Άλλη μια απάντηση πρέπει να βρεθεί. Τρίτον, έρευνα και καινοτομία. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα είναι αποτελεσματικά ή περιορίζουν την έρευνα. Ιδού ερωτήσεις που χρήζουν απαντήσεις. 26 υποψηφιότητες τα τελευταία χρόνια έχουν παραληφθεί για ενεργές ουσίες αλλά υπάρχει μια τάση της μείωσης των ετοιμάτων συμπεριλαμβανομένων και των εναλλακτικών χαμηλού κινδύνου. Έτσι, καμία καινούργια ενεργό ουσία δεν έχει τεθεί προσέγγιση τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Η Μέρη Μακίνες στο τέλος μας λέει τα εξή. Οι γεωργοί χρειάζονται μια πρόσβαση σε πολλά εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες των φυτών. Αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και το σύστημα που ρυθμίζει τα εργαλεία θα πρέπει να είναι επίση αποτελεσματικό, παραγωγικό και διαφανέ, ούτω ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτέ έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και φθηνά τρόφιμα και ότι οι γεωργοί έχουν πρόσβαση σε μέσα παραγωγή αυτών των τροφίμων, χρησιμοποιώντα προϊόντα τα οποία είναι ασφαλή για την υγεία του. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε όλους τους στιώδεις συζητητές. Θα ακούσουμε τώρα τις παρεμβάσεις στο μέλλον της Επιτροπής. Καθώς έχουμε καθυστερήσει λίγο ε, και έχουμε ε, ένα σχετικά μεγάλο αριθμό συναδέλφων που έχουν ζητήσει το λόγο, θα πρέπει να θέσω ένα όριο δύο λεπτών για το χρόνο αγόρευσης. Ε, τη Ράγια, πήρε Πύρεκ λοιπόν ως πρώτη συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τον εισηγητή θα ήθελα να πω πως ε, έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για την γλυφοσάτη και οι πολίτες ε, στην Ολλανδία θέλουν να ξέρουν ξεκάθαρα τι γίνεται ειδικά όσον αφορά τα απορροπαντικά. Και βέβαια το θέμα είναι το θέμα εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα. Αυτά νομίζω έχουν αποδειχτεί ήδη και έχει αποδειχτεί ήδη πολλές φορές πως ανεξάρτητα είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί ειδικά σε σύγκριση με τρίτες χώρες και κάτι άλλο. δεν έχουμε ακόμη καταλήξει και οριστικοποιήσει τι θα γίνει με την αντιμετώπιση των ε, ουσιών εκείνων ε, τα οποία είναι χαμηλού κινδύνου. Δεν είναι δυνατόν να απαγορεύουμε κάτι και μετά να μην υπάρχει καμία λύση. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ περίπλοκη, ακριβή και αργή. Και έχουμε ακριβώς αυτές τις ουσίες χαμηλού κινδύνου, οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν τρόφιμα. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιό να καταλήξει σε κάποια κριτήρια για τις ουσίες ε, χαμηλού κινδύνου. Και τέλος, όταν μιλάμε για το ότι εξαρτώμεθα από τις χώρες για να γίνει κάτι νομίζω ότι κάτι μπορεί να γίνει με τους αγρότες στην Ολλανδία με τα νέα νοικοτινοειδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι με το να απορρίπτουμε κάτι υιοθετούμε το αντίθετό του. Πρέπει κάποια στιγμή να ληφθεί μια απόφαση και να εφαρμόζονται τα όσα αποφασίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία Μελιόρα. Θα ήθελα να πω πως ε, είναι νομίζω μεγάλο πρόβλημα το ότι χάνεται και η εμπιστοσύνη των ε, πολιτών και μεταξύ των αρχών από ό,τι βλέπω και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό είναι καλοδεχούμενη και η πρωτοβουλία διαφάνειας ε, της Κομισιόν. Αν έχουμε λοιπόν ε, έναν καλό κανονισμό, κάτι το οποίο νομίζω επιβεβαιώθηκε και σας ευχαριστώ για την μελέτη η οποία υποβλήθηκε, είναι παρόλα αυτά προβληματικό το ότι διαπιστώνουμε ότι και οι τρεις στόχοι, δηλαδή η υγεία των πολιτών, η προστασία του περιβάλλοντος και το να έχουμε καλά γεωργικά προϊόντα ε, δεν έχουν επιτευχθεί. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να σκεφτούμε το τι συμβαίνει. Και από ό,τι μας δείχνει η μελέτη, κυρίως φταίει η εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να τα έχουμε αυτά όλα κατά νου, να μην αλλάζουμε μόνο τους νόμους, αλλά να κοιτάμε και την εφαρμογή στα κράτη-μέλη λεπτομερώς. Αναφέρθηκαν πάρα πολλά σημεία, ποια αρχή κάνει τι, ε, ποια είναι η εθνική αξιολόγηση, ότι δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση και χάνεται η εμπιστοσύνη. Θέλω να το τονίσω αυτό, η εμπιστοσύνη πρέπει να αποκατασταθεί. Και πρέπει και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τέλος, οι 386 εξαιρέσεις πραγματικά είναι πάρα πολλές, δημιουργούν σοβαρές επιφυλάξεις. Έχουμε επίσης και στην Γερμανία την περίπτωση μιας ε, ουσίας η οποία εξαιρέθηκε. Ε, βεβαίως η εξαίρεση πρέπει να αποτελεί εξαίρεση, όχι τον κανόνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ όταν μιλούσαν οι σκιώδες ηγητές. Είχα μια άλλη συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Νομίζω ότι αναφέρθηκε σε σημαντικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη είναι η διαφάνεια. Για εμένα είναι σημαντικό να έχουμε έναν διαιτητή θα έλεγα τον οποίο εμπιστευόμαστε όλοι, δηλαδή κάποιε είναι ασφαλεί, μπορούμε να τι χρησιμοποιήσουμε, άλλε όχι και πρέπει να τι απογορεύσουμε. Γι' αυτό το λόγο όμω πρέπει να έχουμε πίστη στην διαδικασία και στον ε, διαιτητή. Χρειάζεται λοιπόν διαφάνεια που μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Και το δεύτερο βεβαίω ε, είναι οι εξαιρέσει. Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση για να χρησιμοποιούμε δραστικές ουσίες. Ε, επίσης πάλι εδώ πέρα υπονομεύεται η εμπιστοσύνη στον διαιτητή όπως είπα Τρεις πτυχές λοιπόν είναι σημαντικές για εμένα. Πρώτα απ' όλα το θέμα των δραστικών ουσιών και του συνδυασμού τους. Εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αποφασίζουμε ποιες ουσίες επιτρέπουμε και τα κράτη-μέλη κοιτούν το προϊόν και ίσως και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα ρόλο εδώ ή τουλάχιστον υπάρχει καλύτερη επικοινωνία. Δεύτερον, βεβαίως εάν μιλάμε για βιολογικά, συνθετικά, συμβατικά προϊόντα φυτοπροστασίας, πάντα υπάρχει δυνατότητα κινδύνου στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Δηλαδή, όσο θέλουμε να προστατεύσουμε τις ε, καλλιέργειες, παρεμβαίνουμε στη φύση. Ίσως με πάρα πολύ περιορισμένο τρόπο, αλλά είναι μία παρέμβαση. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούμε χαλκό ή πολύ σκληρά. Πολύ σκληρέ συνθετικέ ουσίε και μετά στην επικοινωνία. Στην γλυφοσάτη είχαμε διάφορε μελέτε, αλλά βεβαίω ήταν ε, τελείω διαφορετικέ και οι εκθέσει. Θέλω να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία για να υπάρχει ακριβώς μια σωστή σύγκριση όλων αυτών. Και αυτά είναι τα βασικά. Μετά κάποια άλλα δευτερεύοντα μικρές χρήσεις για να έχουμε υλικά φυτοπροστασίας και για τις μικρές καλλιέργειες και να σκεφτούμε πώς θα έχουμε μια γρηγορότερη αδειοδότηση για τις εναλλακτικέ για τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου. Νομίζω έτσι θα πάει η γεωργία προς ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος ήταν σκιώδης ηγητής τη Άλντε, τον άφησα να μιλήσει λίγο παραπάνω. Θα ήθελα να παρακαλέσω όμω του υπόλοιπου ομιλητέ να περιοριστούν στα δύο λεπτά. Η κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς το EPRS για τη δουλειά που έκανε. Πολύ ενδιαφέρουσα η εργασία. Τώρα σαν αφορά τη διαδικασία θέλω να πω κάτι της εγκρίσεως των δραστικών ουσιών είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η έναρξη. Και μετά πάμε σε όλα τα άλλα. Να υπογραμμίσω το εξή στον κανονισμό. Υπάρχει ένα κενό. Το άρθρο 6, εδάφιο F. Τι λέει εκεί. Ότι είναι οι όροι και οι περιορισμοί. Αν λείπουν πληροφορίες, λέει, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν αργότερα το πρόβλημα αυτό των, της ελλείψεως των στοιχείων των βιομηχανιών είναι κάτι που μπορεί να έχει συνέπειες για την υγεία και το περιβάλλον. Και αυτό είναι ένα κενό του συστήματος κατά την άποψή μου όσον αφορά την ε, έγκριση δραστικών ουσιών. Μετά από κάποια χρόνια, δύο-τέσσερα χρόνια, διότι οι βιομηχανίες δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία, ε, μετά περιορίζουμε την χρήση αυτό σημαίνει ότι δεν εφαρμόζουμε την αρχή της πρόληψης, αλλά είμαστε στην αξιολόγηση του κινδύνου και δίνουμε πολύ μεγάλη ελευθερία στη βιομηχανία για να δώσει τα στοιχεία που λείπουν για την αξιολόγηση της ουσίας. Εγώ θα πήγαινα πιο πέρα. Να πω ότι όσο δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία τοξικολογίας, όλα τα στοιχεία δεν πρέπει να εγκρίνεται η ουσία από τη στιγμή που υπάρχουν τα στοιχεία όλα να γίνεται έγκριση. Διότι βρίσκουμε τις συνέπειες μετά στα κράτη-μέλη. Διότι τα κράτη-μέλη, όπως είπατε, δεν έχουν τις αρμοδιότητες απαραίτητα και κυρίως τον έλεγχο της χρήσεως και αντιλαμβανόμαστε ότι καμιά φορά δέκα χρόνια αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί λάθος οι ουσίες. Αν θέλουν προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων πραγματικά, θα έπρεπε ανάντι να αλλάξουμε κάπως τον κανονισμό όσον αφορά τα κενά των δεδομένων η έγκριση να μην γίνεται παρά μόνο όταν υπάρχουν όλα τα στοιχεία από τη βιομηχανία και σε επίπεδο κρατών μελών να ενισχύσουμε τον έλεγχο ε, όσον αφορά τη χρήση. Ευχαριστώ. Ο κ. Πιέρα είναι ο επόμενο που έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Το θέμα αυτό είναι Πολύ ευρύ. Ε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, ομάδα ε, της Υπηρεσίας Μερωτών του Κοινοβουλίου και τον συζητή μας για αυτά τα σχόλια. Ε, Δυστυχώ, ο συγκεκριμένο κανονισμό δείχνει πολύ καλό σε επιχάρτο, αλλά η εφαρμογή του σε καμία περίπτωση δεν είναι ιδανική. παρά τι διαφορές διαφορέ που παρατηρούμε μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, θεωρούμε πω οι προτεραιότητε του κανονισμού δεν θα πρέπει να μεταβληθούν η συζήτηση την οποία κάνουμε αποτελεί προϊόν μιας άλλης συζήτηση ε, που έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα και η οποία σχετίζεται ακριβώς με την αβεβαιότητα η οποία σχετίζεται με ε, που έχει προκύψει από κάποια περίεργα δημοσιεύματα, κάποιες ε, μελέτες, αλλά και από μια σειρά από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν ε, αυτή η αβεβαιότητα είναι που δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα και νομίζω πως ε, θα πρέπει να τονίσουμε τα κενά που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού, υπογραμμίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι υποστηρίζουμε την κατανομή ε, των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών μεταξύ θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, κρατών μελών, αλλά ε, και αγροτών, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά τους και γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες ε, τόσο του κλάδου τους όσο και του περιβάλλοντος. Οπότε δεν θα πρέπει να τους επιβληθούν σε αυτούς τους αγρότες διατάξεις άνωθεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτές και αυτό αποτελεί ένα ζήτημα κέρια σημασία και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε και τόσα πολλά προβλήματα στο επίπεδο τη εφαρμογή. Ευχαριστώ, λέω. Ο πρόεδρο, κύριε Νταλή, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κατά τελευταία χρόνια έχουμε κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα συζήτηση για αυτό το ζήτημα και ειδικότερα για τη γλυφοζάτη. Ε, ο συνάδελφός μου αναφέρθηκε μόλις τώρα και στο ζήτημα της έλλειψης εμπιστοσύνης στο σύστημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αν δούμε τα απορίσματα από ορισμένε επιστημονικές μελέτες τα οποία καταδεικνύουν ότι ορισμένες από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι καρκινογόνες και κατά συνέπεια ε, μπορούν να έχουν συνέπειες ε, για την ανθρώπινη υγεία, για παράδειγμα και ενδοκρινικοί διαταράκτες οι οποίοι δηλαδή μπορούν να διαταράξουν το ενδοκρινικό σύστημα, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και είναι υποχρέωσή μας να φροντίσουμε έτσι ώστε οι δραστικές ουσίες τις οποίες εγκρίνουμε να μην έχουν αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία το περιβάλλον και την υγεία των ζώων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί πραγματικά πιστεύω ότι έδειξε ότι η δική μας Επιτροπή έχει αναλάβει την ευθύνη να συνεχίσει τη συζήτηση αυτό το ζήτημα και θέλει να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση των ε, φυτοπροστατευτικών ε, προϊόντων. Εάν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ε, καλή νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην εναρμόνιση των διατάξεων, αλλά και στον τρόπο παρακολούθηση των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στι καλλιέργειε τη ευρωπαϊκή αγορά. Η εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και η εναρμόνιση μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών και ε, διατάξεων και μάλιστα η έλλειψη που υπάρχει σήμερα οδηγεί σε έλλειψη σε ό,τι αφορά τα κατάλληλα δεδομένα, πράγμα το οποίο αποτελεί με τη σειρά του πρόβλημα για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Άρα λοιπόν μια κοινή πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μας έδινε περισσότερη ορατότητα σε ό,τι αφορά ε, την, ε, και τα οικονομικά δεδομένα αλλά και την χρήση άλλων εναλλακτικών. Ωστόσο, για να επιτευχθούν όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει και ε, και πρόσβαση σε εναλλακτικέ. Κατά τη συνέπεια, νομίζω πω είναι σημαντικό να προωθήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Λόρεντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. με αυτά που ακούω εδώ πέρα, πραγματικά εκπλήσω με το ότι ζούμε ακόμα, βρισκόμαστε εν ζωή. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, χρησιμοποιώ ως αγρότης ε, και φυτοφάρμακα ε, εγώ τα χρησιμοποιώ αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, ε, άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο αναφέρει ο κ. Πότσα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσει στον κανονισμό και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε η συζήτηση σε ό,τι αφορά τα νέο νοικοτινοειδή κατέδειξε ότι γνωρίζουμε πολλά σε ό,τι αφορά το νερό, αλλά πολύ λίγα σε σχέση με το έδαφος. Και τώρα βλέπουμε ε, τα δείγματα τα οποία λαμβάνονται από διάφορες διαφορετικές ε, καλλιέργειες και βλέπουμε ότι υπάρχουν φυτοφάρμακα σε τέτοιου είδους εδάφη τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε τέτοιου είδους ε, καλλιέργειες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναλάβουμε δράση και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των εξαιρέσεων θα συμφωνήσω πλήρως με τον συνάδελφο από τους πράσινους. Δηλαδή οι εξαιρέσεις θα πρέπει να ισχύουν σε ελάχιστε περιπτώσει και θα πρέπει να καταρτήσουμε ενδεχομένω ε, και ένα θετικό κατάλογο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί με βάση το σημερινό θετικό κατάλογο έχουμε ε, κράτη-μέλη τα οποία λαμβάνουν 800 ή 1000 προϊόντα από αυτού, ενώ άλλα κράτη-μέλη τα οποία λαμβάνουν μόνο 20 προϊόντα. Οπότε υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ό,τι αφορά την επιλογή που κάνουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Και εδώ έρχομαι σε κάτι που ανέφεραν και οι φιλελεύθεροι. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά κάποια, για παράδειγμα, φρούτα του δάσου, ε, βατόμουρα για παράδειγμα ή άλλα, έχουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά τις, ε, την αναφορά τις αναφορές που δεν έχουν τα, τα, κατάλληλα δεδομένα και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτό το τομέα τα γνωρίζουν. Οπότε θα πρέπει να αποφύγουμε την εισαγωγή προϊόντων τα, στα οποία χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα τα οποία εμεί δεν επιτρέπουμε. Θα πρέπει σε κάθε λοιπόν περίπτωση να συνεχίσουμε τι βελτιώσει σε αυτόν τον κανονισμό σε ό,τι αφορά τι εγκρίσει, αλλά δεν νομίζω πω ε, απλώ ε, και μόνο η Επιτροπή ΠΕΣ μπορεί να επιτύχει κάτι εδώ. Θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω υποστήριξη για αυτή την εργασία και θα πρέπει να συνεχίσουμε εδώ τι εργασίε μα. Ευχαριστώ κύριο Στάσα, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για να απαντήσω στον Καλχάιντ Φλόρεντς. Ναι, όλοι ζούμε Πράγματι, αλλά μελέτες στη Γερμανία δείχνουν ότι 75% των εντόμων έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχει λοιπόν σοβαρός αντίκτυπος ε, στο περιβάλλον. Ευχαριστώ λοιπόν την υπηρεσία μελέτης. Ε, και στο 1,5 ε, λεπτό που μου απομένει θα ήθελα να επικεντρωθώ στις εξαιρέσεις ε, που αναφέρθηκε στην παράγραφο 17 και 18 στην 17 ζητάμε να περιορίσουν τα κράτη-μέλη της εξαιρέσεις. στο άρθρο 53 της ε, σχετικής ε, οδηγίας βλέπουμε εδώ πέρα πως και η Κομισιόν έχει ένα ρόλο να παίξει μπορεί να πάει στην ΕΦΣΑ, μπορεί να πάει στην μόνιμη επιτροπή πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τον ρόλο της Κομισιόν και θα ήθελα να ρωτήσω την ε, Κομισιόν πώς βλέπει τον ε, ρόλο της εδώ πέρα θεωρεί ότι είναι επαρκώς ε, ενεργή. Στην παράγραφο 18 ακριβώς μιλάμε για το πώς υπάρχει η προσαρμογή των διαφόρων μεθόδων. Και ακριβώς ε, το ερώτημα είναι τι κάνετε για να εφαρμοστούν αυτά, τι κάνετε στην επιτροπολογία και οι μέθοδοι που ακολουθούνται αν μπορείτε να μας πείτε κάποια περισσότερα για αυτές. Ευχαριστώ κυρία Ρίς. Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω το EPRS για την εξαντλητική αυτή ανάλυση που έκανε. Και από τη συζήτηση βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές και δυσλειτουργίες όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού. Και αυτό δικαιολογεί τις εργασίες μας στην έκθεση του κ. Πορτ και το έργο της Επιτροπής. Κυρία Καραμφίλοβα, η κυρία Καραμφίλοβα ξεκαθάρισε τα πράγματα την αρχή και είπε στην αρχή ότι κανένας από τους στόχους, κανείς από τους στόχους του κανονισμού δεν επετεύχθη. Αυτό είναι πολύ ευστηρό όσον αφορά την υγεία εσωτερική αγορά, παραγωγή γεωρικών προϊόντων από την αρχή ε, στη μελέτη. Βλέπουμε ότι όλοι οι φορείς, η παραγωγή, οι καλλιεργητές, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι εθνικές αρχές Όλοι συμφωνούν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η λήψη αποφάσεων λαμβάνεται με τον καλύτερο τρόπο. Άρα ξαναθέτω το ερώτημα. Δεν έχω πολύ χρόνο. Να θέσουμε το ερώτημα ξανά. Θα πρέπει ίσως να εξετάσουμε τη δυνατότητα να λήξει αυτό το διτό σύστημα που είναι ακρογωνιω λήθος της λήψης αποφάσεων. Δηλαδή αξιολόγηση και έγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ουσία και σε επίπεδο κρατών μελών όσον αφορά το προϊόν. Βασικό ερώτημα απηχεί και το πρώτο ερώτημα της έξοχης εκθέσεως του εισηγητού ε, και εγώ συμφωνώ με τις περισσότερες διαπιστώσεις και συστάσεις. Να επιμείνω επί δύο σημείων που ήδη αναφέρθηκαν. Καταχρηστική προσφυγή στην κατεπίγουσα διαδικασία στο σημείο 4 και 17 της έκθεσης αναφέρεται πρέπει να τεθεί τέρμα στην κατάχρηση των εξαιρέσεων που δικαιολογούνται από το άρθρο 53 που δικαιολογεί περιστάσεις ειδικέ. Ειδικέ ε, είναι πολύ αόριστο και βλέπουμε ότι που οι καταπήγουσε δικασίε σε συνέχεια παρατείνονται, παρατείνονται και φτάνουν σε διαδικασίε που δεν έχουν τίποτα, καμία σχέση με το κατεπήγον. Θα το τροποποιούσα και το άλλο. Το παράρτημα που προβλέπετε για τον αρνητικό, κατά... κατάλογο, δέκα χρόνια παραμένει κενό ο κατάλογος μετά τον κανονισμό. Για τα υπόλοιπα, συμφωνώ με τα συμπεράσματα της εκθέσεως του κυρίου Ποκ. Ευχαριστώ. Επόμενος, ο κ. Αντριού, πρόεδρος Επιτροπής ΠΕΣΤ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω το EPRS για την εργασία που έκανε και ευχαριστώ και τον Πάβελ. Καταδεικνύει ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα σήμερα και επίκαιρο. Οι περισσότεροι που μίλησαν με οδήγησαν σε προβληματισμό. Χρειάζεται δουλειά κοινό διακύβευμα, η ανθρώπινη υγεία, στο και των ησυχιών μας. Μπορούμε να θεσπίσουμε την καλύτερη δυνατή νομοθεσία, μπορεί να έχουμε το... Λοιπόν, έχουμε διάφορα προβλήματα με το προστάτη και στους καρκίνους δεν μπορούμε, τέλο του έχουν εξαφανιστεί διάφορα έντομα και διάφορα πτηνά κλπ. Και δεν μπορούμε να κάνουμε επίσης ότι ε, δεν τρέχει τίποτα. Και με τις μέλισσες υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό διαδηλώνουν οι μελισσοκόμοι σήμερα. Διότι ε, τα έντομα αυτά που βοηθούν στην επικονίαση των ε, φυτών εξαφανίζονται. Λοιπόν, η μελέτη πρέπει να μας οδηγήσει σε προτάσεις συγκεκριμένες στην Επιτροπή ΠΕΣΤ για να καλύψουμε τα διάφορα κενά που υπάρχουν υπάρχουν διάφορα προς βελτίωση. Είμαστε υπεύθυνοι εμείς, πολύ υπεύθυνοι ε, για την βελτίωση της αδειοδότησης των παρασιτοκτόνων. Δεν έχουμε χρόνο που σε λεπτομέρειες. Δηλαδή τι γίνεται από την έρευνα, ποια μέσα τη θέτει, ποια είναι η θέση της βιομηχανίας σχέση με την έρευνα. Των δύο επιπέδων του ευρωπαϊκού και του εθνικού σαν αδειοδότηση θα έχουμε διάφορε προτάσει συγκεκριμένε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση τη νομοθεσία. Αυτό ισχύει για το μέλλον τη Γεωργία. Πρέπει να το αντιληφθούμε διαφορετικά ε, για, για τα γεωπονικά θέματα και για την ανθρώπινη ε, υγεία των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Ε, και θα πρέπει να πετύχουμε τους στόχους μα. Αυτή είναι η αποστολή μα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάλενμπαχ. Ευχαριστώ πολύ και για την επιστημονική επεξεργασία του θέματος και για την πρόταση του κυρίου Πότς. Θεωρώ ότι το τωρινό ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης και βεβαίως χαιρετίζω την πρωτοβουλία να επανεξεταστεί για να έχουμε ένα αποτελεσματικό και αποτελεσματικό σύστημα αδειοδότησης που θα βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου. Συνοψίζοντας όσα ακούστηκαν, θα έλεγα ότι ως Επιτροπή Περιβάλλοντος πρέπει να προσέξουμε τη μελλοντική αγροτική πολιτική να παίξουμε έναν σημαντικό ρόλο. Το θέμα δεν είναι μόνο η αδειοδότηση και η διαφάνεια, αλλά και το ποιες ποσότητες ε, χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, δηλαδή ε, για να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν λιγότερα ζυζανιοκτώνα για να μειωθεί ο κίνδυνος για άνθρωπο και περιβάλλον. Αυτά τα οποία λέγαμε. Δηλαδή μια ευρωπαϊκή γεωργία που θα είναι ανταγωνιστική θα παράγει τρόφιμα και ζωοτροφές σε αποτελεσματικό επίπεδο και αυτό δεν θα γίνει ποτέ χωρίς ε, ζυζανιοκτώνα, αλλά υπάρχουν νέα ζυζανιοκτώνα, βιολογικά, άλλες μορφές καλλιέργειας που πρέπει να αναπτύξουμε και βεβαίω γι' αυτό χρειάζονται και τα απαραίτητα κονδύλια, αναφέρθηκαν οι επενδύσεις στην έρευνα. Η δεύτερη αποστολή είναι η καλύτερη νομοθεσία, η οποία όσο καλή και να είναι δεν χρησιμεύει τίποτα εάν δεν εφαρμόζεται. Και αυτό δεν είναι μόνο δουλειά της ε, Κομισιόν αλλά και των ε, βουλευτών σε συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί εδώ υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλές εξαιρέσεις ε, σύμφωνα με το άρθρο 53 για να το συζητήσουμε και στα διάφορα κοινοβούλια. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι και στο μέλλον με την νομοθεσία αυτή θα επιτύχουμε τους στόχους που δεν έχουμε ακόμα πετύχει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ε, μπορείτε να στείλετε γραπτός στην υπηρεσία έρευνας. Να δώσω τώρα τον λόγο στην Κομισιόν στον κύριο Μπέρεντ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την υπηρεσία, ευχαριστώ και τον κύριο Πότς για την έκθεση και για όσους μίλησαν για τα θέματα αυτά. Κοιτάξτε, νομίζω τα ευρήματα της έκθεσης αυτή συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τα όσα διαπιστώσαμε στην μελέτη που προετοιμάστηκε για την Κομισιόν στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης της ε, νομοθεσίας ε, και βεβαίως η ειδική αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό η ίδια, οπότε δεν προξενεί έκπληξη αυτό και τα ευρήματα συμφωνούν με τα όσα βρίσκουν οι επιθεωρητές ε, στους επιτόπιους ελέγχους στα κράτη-μέλη. Να ξεκινήσω με κάποια από τα θετικά, ότι ο κανονισμός θεωρείται πραγματικά σχετικός και σημαντικός για τις πραγματικές ανάγκες. Με εξέπληξε λίγο αυτό το οποίο λέει η υπηρεσία έρευνα ότι κανένα στόχο δεν έχει επιτευχθεί γιατί αυτό το οποίο περιγράφει μετά η έκθεση είναι κάπω ε, πιο διαφορετικό. Παραδείγματο χάρη, η ίδια η έκθεση λέει ότι οι ενδιαφερόμενοι όλων των κατηγοριών συμφωνούν ότι οι περιβαλλοντικοί στέχοι έχουν επιτευχθεί εκτός από τις ε, ΜΚΟ και τον κλάδο των ε, βιολογικών ζυζανιοκτώνων. Κάτι ανάλογο βρήκαμε και εμεί για τις άλλε απόψει, ανταγωνιστικότητα κτλ. Επίσης είναι διχασμένες οι αποψει οπότε ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, είναι κάπως ε, διαφορετική η κατάσταση, έχει αποχρωσει Και επίσης ε, για την γλυφοσάτη αναφέρει η έκθεση της EPRS ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για λανθασμένο χειρισμό. Τώρα για αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Πότς και πολλοί από τους κοιόδης εισηγητές εδώ η Κομισιόν συμφωνεί με πολλούς από αυτούς ειδικά στις καθυστερήσεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη δεν γίνονται σεβαστές οι προθεσμίες για αξιολογήσεις. Ε, ανησυχούμε πάρα πολύ με αυτό και αυτός είναι ο λόγος για τα περισσότερα προβλήματα τα οποία σχολιάστηκαν και προκύπτουν από αυτά. Ειδικά η κατάχρηση του άρθρου 53 για εξαιρέσεις είναι άμεση συνέπεια των καθυστερήσεων και το ότι δεν υπάρχει το σύστημα αμοιβαία αναγνώριση. Ε, τα κράτη-μέλη δεν εμπιστεύονται αλλήλους. Τούτου λεχθέντος ε, η έκθεση σημειώνει και το επιβεβαιώνουν και τα ευρήματά μας ότι 90% των εξαιρέσεων είναι για προϊόντα που περιέχουν ουσίε που είναι εγκεκριμένε. Δεν είναι για ουσίες που δεν είναι εγκεκριμένε. Οπότε αν τα κράτη-μέλη αξιολογούσαν τα προϊόντα στην κανονική διαδικασία δεν θα χρειαζόταν την διαδικασία του άρθρου 53. Ο κύριος Στάς συγκεκριμένα ρώτησε τι κάνει η Κομισιόν. Ζητήσαμε από την Εύσα να αξιολογήσει πέρσι το εάν οι εξαιρέσει που δόθηκαν για τα νέο νοικοτινοειδή που είχαν περιοριστεί πέρσι ήταν δικαιολογημένε ή όχι. Και η ΕΦΣΑ μόλις οριστικοποίησε την απάντησή της, ε, την εξετάζουμε. Μπορώ να σας πω προκαταρκτικά το εξής, ότι για αρκετά για αρκετούς συνδυασμούς ε, φυτών και ζυζανίων ε, δεν υπήρχαν εναλλακτικέ. Για άλλους υπήρχαν, οπότε δεν θα έπρεπε να έχουν δοθεί εξαιρέσεις. Τώρα, ο κανονισμός μας δίνει την δυνατότητα να δοθεί κάποια συνέχεια με αποφάσεις της Κομισιόν. Εξετάζουμε τις ε, περιπτώσεις αυτές ε, Ο κύριος Στάς επίσης ρώτησε για το αν χρειάζεται περισσότερη κατεύθυνση για τις ε, δυνατότητες ε, αξιολόγησης του κινδύνου με βάση τα κριτήρια για τα όρια για το άρθρο 7. Πράγματι προσπαθούμε να συμφωνήσουμε με τα κράτη-μέλη για το τι είναι η αμεληταία έκθεση. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταφέρει αλλά συνεχίζεται η δουλειά και η ΕΦΣΑ έχει αναπτύξει ένα ξεκαθαρό πρωτόκολλο για το πώς τα κράτη-μέλη πρέπει να αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάγκη φυτογειονομική και ισχύει το άρθρο 7 για τις ε, αδειοδοτήσεις αυτές εκτακτού ανάγκης. Ε, κάποια άλλα σημεία που αναφέρθηκαν ε, είναι το ότι διαφέρνει οι ικανότητες στα κράτη-μέλη και οι πόροι. Είναι σαφές ότι δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να κάνουν τις αξιολογήσεις, αλλά και πάλι αυτό αντισταθμίζεται από τις ε, τους ελέγχους και από τον έλεγχο της ΕΦΣΑ αλλά όπω είπαμε στα προϊόντα αυτοποστασίας δεν είμαστε ακόμα εκεί που πρέπει να είμαστε. Πολλοί σχολίασαν για τη διαφάνεια, την έλλειψη διαφάνεια και σημείωσαν επίση ότι οι προτάσει τη Κομισιόν για την τροποποίηση του, κανονισμού, του Γενικού Κανονισμού για τα Τρόφιμα ήδη αναφέρθηκε σε κάποια από αυτά τα σημεία και πράγματι θεωρούμε ότι οι προτάσεις αυτές θα βοηθήσουν την αύξηση της διαφάνειας. Ο κύριος Πότς πρότεινε επίσης να το σκεφτούμε αυτό στην φάση της διαχείρισης του κινδύνου και το σημείωσα. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι για τις πιο δύσκολες όπως η γλυφοσάτη και τα νεονικοτινοειδή έχουμε συγκεκριμένα site όπου αναφέρουμε αμέσως ότι γίνεται στις συζητήσεις στην Επιτροπή ποιες είναι οι προτάσεις μας. Αυτό λοιπόν μπορεί ίσως να ακολουθηθεί και για άλλες ουσίες ε, στο μέλλον και θα το σκεφτούμε. Πολλοί ομιλητές επίσης ανέφεραν ε, τη διαδικασία των επιβεβαιωτικών δεδομένων. Εδώ πέρα θεωρούμε ότι η Κομισιόν σέβεται τους ε, κανόνες ε, στον κανονισμό. Η κυρία Ριβαζή επίσης το ανέφερε. Υπάρχουν δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα, η διαδικασία αυτή. Υπό όρους δεν είναι βεβαίως μία εξουδότηση λευκό και το έχουμε παραπέμψει το θέμα στον διαμεσολαβητή. Εμείς θεωρούμε ότι ευθυγραμμιζόμαστε με τους όρους ε, του κανονισμού. Συνοψίζοντας λοιπόν, συμφωνούμε με την εντύπωση όσων ε, λένε ότι έχουμε ένα πολύ αυστηρό καθεστώς, ίσως το αυστηρότερο στον κόσμο. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση στην εφαρμογή. Και βεβαίω οι κύριοι δρόντε εδώ είναι τα κράτη-μέλη. Οπότε αναμένουμε τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και οπωσδήποτε θα τα λάβουμε αυτά υπόψη όταν θα οριστικοποιήσουμε την δική μας αξιολόγηση και θα σκεφτούμε τα επόμενα μελλοντικά βήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λόγω στον κύριο ποτ, θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομο γίνεται. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του για αυτά που είπαν και για τη συνεργασία μέχρι τώρα και προσβλέπω στη συνέχιση αυτής. Μπορούμε τώρα πια να εκπληρώσουμε το ρόλο μας. Μετά τη συζήτηση να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις στο μέλλον. Λυπούμε που η κυρία Μίλλερ δεν είναι εδώ πια. Για να πω κάτι ξεκάθαρα, ποτέ δεν επέκρινα τον κανονισμό αυτό κάθε αυτό. Δεν είναι ρόλος μου. Δεν το έκανα στην έκθεσή μου ούτε στην παρέμβασή μου. Κάποια παρεξήγηση έγινε. Το καλύτερο εργαλείο για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, λέω. Ε, έτσι αναφέρω τον κανονισμό. Θέλω να βελτιωθούν τα τμήματα του κανονισμού και της υλοποίησης αυτού που χρειάζεται. Για τον κάλ τον συνάδελφο, μη φοβάστε, δεν προσπαθώ να παρουσιάσω σκοτεινές εικόνες. Σέβομαι την έρευνα της Ευρωπαϊκής, της ε, υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, της υπηρεσίας έρευνας του Κοινοβουλίου. μπορώ να σας στείλω για κάθε δήλωση της εκθέσεώς μου παραπομπές από την έρευνα. Αυτή η έκθεση και η δουλειά μας αφορούν την βελτίωση της εφαρμογής. Δεν θέλουμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία αυτή καθε αυτή, αλλά την εφαρμογή της. Αυτός είναι ο ρόλος της Επιτροπής ΠΕΣΤ, και όχι της εκθέσεως αυτής. Είπα ότι περιμένω ότι η δική μας ε, υπηρεσία έρευνας ε, λειτουργεί πολύ καλά. said about Όταν ικανοποιημένοι εμπλεκόμενοι φορείς με την εφαρμογή κάποιας νομοθεσίας, αυτό δεν είναι απαραίτητα ένα μήνυμα ότι εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία. Αυτό είναι τα αστιακή μου. Ευχαριστώ. Και προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση επί του θέματος. Χρονοδιάγραμμα για τροπολογίες. Προθεσμία 12 Ιουνίου στις 11 η ώρα ψηφοφορία ενδεχομένως τον Ιούλιο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην Ολομέλεια ε, δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Επόμενο σημείο. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την, την οδηγία για τα θέματα υγείας, αξιολόγησης, την τοπολογία του κανονισμού. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον εισηγητή όσον αφορά την τεχνολογία υγείας. Θα ξεκινήσω, Πρόεδρε, λέγοντας ότι η πρωτοβουλία μου φαίνεται ότι είναι ενδιαφέρουσα και μπορεί να ενισχυθεί η Ευρώπη να κατα... και να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντική αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγεία και αυτή η πρόταση προχωρεί προς την κατεύθυνση. Βέβαια υπάρχουν και διάφορες δυσκολίες όσον αφορά την, ε, τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το θέμα της υγείας ε, των ασθενών, να βελτιώσουμε την πρόσβαση της τεχνολογία όσον αφορά την υγεία. Γι' αυτό είμαι πεπισμένη. Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδου σημασία λοιπόν αυτή η πρόταση να παράγει επαρκή ε, εμπιστοσύνη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να γίνεται ποιοτική δουλειά, να επικρατεί διαφάνεια, να υπάρχει ανεξαρτησία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε μέσω των τροπολογιών που έχω υποβάλει. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του για την πρόσβαση στα φάρμακα και στην περίθαλψη πέρσι θέλει μία εναρμόνιση όσον αφορά την τεχνολογία της υγείας και τη διαγνωστική. Και πιστεύω ότι αυτό είναι θεμελιώδες βήμα για τη βελτίωση της, της ποιότητας της έρευνας. Πρέπει να, ε, να έχουμε κλινική ε, αξία όσον αφορά των ιατρικών αυτών τεχνολογιών, να βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών σε αυτή τη τεχνολογία για την υγεία και να έχουμε σωστέ προτεραιότητε για την καινοτομία. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη, βασίζεται στη λειτουργία τη εσωτερική αγορά, η οποία στον τομέα είναι κατακαιρματισμένη. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι το βασικό πρόβλημα και δεν είναι και το μοναδικό πρόβλημα. Αυτή η πρόταση θα μπορούσε να επικεντρωθεί επί των διαφόρων στόχων που έχω παρουσιάσει και τη βελτίωση της ενίας αγοράς μεταξύ άλλων. Οι βασικές αλλαγές έχουν σαν στόχο ε, μια επιστημονική αξιολόγηση. Επιστημονική αξιολόγηση υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιεί το μέγιστο αριθμό των κλινικών στοιχείων και αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται από εμπειρογνώμονες που είναι ανεξάρτητοι από εθνικού φορεί ε, αξιολόγηση των ιατρικών τεχνολογιών. Θα πρέπει να είναι αξιολόγηση σε επιστημονικές διαφανείς, αντικειμενικές και γι' αυτό το λόγο έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό στόχο. Δηλαδή θα πρέπει η μεθοδολογία που εφαρμόζεται να είναι διαφανής, αντικειμενική, υψηλή ποιότητα, και θα πρέπει να προωθείται από εμπειρογνώμονε οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και δεν δέχονται κάποιε επιρροέ και παρεμβάσει. Χρειάζεται μεθοδολογία αρκετά ευέλικτη ούτω ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ε, στη χρήση των περισσότερων στοιχείων για την αξιολόγηση. Θα πρέπει οι εγκρίσεις να γίνονται ε, με μεγαλύτερη πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάνω από τα δύο τρίτα, για να δοθεί μεγαλύτερη δύναμη στι αποφάσει, αλλά πρέπει να υπάρχει και ισορροπημένη συμμετοχή, δημοκρατική συμμετοχή των κρατών μελών ε, που καλούνται να συμμετάσχουν. Πρέπει να χρησιμοποιούνται επιστημονικά κριτήρια και όχι πολιτικά κριτήρια. Δύο τρίτα στις ψήφους και μετά υποχρεωτική αξιολόγηση. Αυτό είναι και το πιο επίμαχο σημείο που αφορά τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να πεθυμίσω τρεις φάσεις της συνεργασίας θελοντικής μέχρι τώρα δεν ήταν επιτυχής, δεν οδήγησαν συνοθέτηση της εκθέσης. πρέπει να εγγυηθούμε λοιπόν να υπάρξει αυτός ο μηχανισμός και να λειτουργήσει. Όταν θα υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη είναι πιθανόν χάρη σε μια διαδικασία υψηλής ποιότητας επιστημονικής να μην χρειάζεται ε, να εφαρμόζονται τα διάφορα μέτρα. Θα πρέπει όμως να υπάρχει εγγύηση ότι θα λειτουργεί σωστά αυτός ο μηχανισμός, να ξεκινήσει να λειτουργεί. Είμαι πεπισμένη ότι με τις ε, τροπολογίες, σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη-μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους όσον αφορά τη κλινική αντιμετώπιση και με δικαιολογημένο τρόπο μπορούμε να οδηγηθούμε σε άλλη αξιολόγηση βάσει ειδικών χαρακτηριστικών. Αυτή είναι μια από τροπολογίες που υποβάλλω. Πιστεύω ότι έτσι σεβόμεθα την διαδικασία λήψη αποφάσεων των μελών. Πεδίο εφαρμογή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει αυτή η κεντρική αδειοδότηση για τα φάρμακα υψηλού κινδύνου και για τους διάφορους ιατρικούς μηχανισμούς. Κατά την άποψή μου πρέπει να βασιστούμε κυρίως επί της καινοτομίας, της πιο σημαντικής καινοτομίας που έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο για τη δημόσια υγεία. Πιστεύω επίσης και για τον, ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο του οικονομικό. Ποιε είναι οι καινοτομίε, ποιε είναι οι νέε τεχνολογίε, ποιε είναι αυτέ που καλύπτουν κενά. Όταν τα ιατρικά, ιατρικές συσκευές όσον αφορά αυτό το θέμα συζητείται είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον συμπεριφθεί στην πρόταση, διότι αυτή είναι μια αγορά ιδιαίτερα ε, ενδιαφέρουσα. Υποσχέται πολλά περισσότερα από τα φάρμακα και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να ε, καλυφθούν τα διάφορα κενά που υπάρχουν όσον αφορά τα στοιχεία και που εμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων. Ε, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου για την ασφάλεια, αλλά πρέπει να κάνουμε σημαντικά βήματα πρόοδου για κατανοώντας την προστιθέμενη αξία τη θεραπευτική, ποια είναι το ωφέλη. Αυτό είναι σημαντικό και για την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη. Να πετυχάνουμε προστιθέμενη αξία χάρη σε αυτό το πιστοποιητικό, αυτό το σήμα ποιότητα που μπορεί να δώσει η αξιολόγηση. Θα πρέπει λοιπόν, κατά την άποψή μα, συμπεριλάβουμε και αυτό το στοιχείο και θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι ίσω μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτά τα μηχανήματα ή αυτέ τι τεχνολογίε που καλύπτουν κενά ή που έχουν αντίκτυπο για τη δημόσια υγεία. Πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο ταυτόχρονα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή για το θελοντικό σύστημα και εδώ μπορούν τα πράγματα. Μπορούμε να, να δούμε τα, την ακριβή ιατρική που απαιτεί νέε μεθοδολογίε, νέε διαδικασίε. Όχι μόνο την, ε, να μην επενδύουμε σε απειρχιόμες τεχνολογίε, να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών ε, και διάφορου συνοδευτική θεραπεία κλπ. Παρηγορητική θεραπεία κλπ. Λοιπόν, Όλα αυτά είναι τα στοιχεία για την εθελοντική εφαρμογή. Όσον αφορά το διάλογο, είναι σημαντικός για τη βελτίωση αποτελεσματικότητα και την πρόθεση της έρευνα και έχω υποβάλει σχετικέ τροπολογίε. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι θεμελιώδης ο ρόλος της. Θα πρέπει να υποστηρίξει τις προσπάθειες. Γι' αυτό ζητούμε στην έκθεση η χρηματοδότηση να γίνεται από το δημόσιο τομέα και να προέρχεται τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να εγγυηθούμε έτσι την ανεξαρτησία. Λοιπόν, θα πρέπει να επικεντρωθούμε επί του ασθενούς και πιστεύω ότι είναι αδύνατο να πετύχουμε συμφωνία διότι πρέπει να θυμηθούμε πάντα ότι βασικός δικαιούχος θα πρέπει να είναι ο ασθενής. Τώρα επικουρικότητα. Η πρόταση με τις τροπολογίες που υπευλήθησαν ε, σέβεται σαφώς την επικουρικότητα κυρίως υπενθυμίζοντας ότι εδράζεται ουσιαστικά επί επιστημονικής αξιολογήσεως που είναι αντικειμενική από πλευράς κλινικής, κλινικών ερευνών. Δεν υπάρχει κάποια επιρροή και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τις εθνικές αρμοδιότητες. Πιστεύω ότι αυτό είναι χρήσιμο ούτως ώστε να καθορίζονται και τιμές αποζημίωσης αλλά δεν θα πρέπει να στραφούμε κατά τη αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών επ' αυτού. Εν γέννη, η πρόταση είναι καλή. Ε, αποτελεί μια ευκαιρία και όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα, έχουμε αναφερθεί σε διάφορε διατάξει για τη βελτίωση τη πρόσβαση στα φάρμακα για του Ευρωπαίου πολίτε. Σε διάφορου τομεί είναι απαραίτητο να κάνουμε προσπάθειε, αλλά το βασικό είναι το εξή. Θα πρέπει να βρούμε μια συμφωνία, θα πρέπει να συνεργαστούμε αυτή η πρόταση έχει αυτό το στόχο και πιστεύω ότι είναι θετική και πρέπει να υποστηριχθεί. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Καθώς είναι πολύ περιορισμένο το χρονοδιάγραμμα μας, ε, θα περιορίσω το χρόνο ακόμη των σχεδόν σε τρία λεπτά και των υπολείπων ε, συναδέλφων σε δύο λεπτά. Ε, η κυρία Χάλια Πύρεκ, λοιπόν, ως συγγήτρια για το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Εκπροσωπώ την κυρία Γκροστέτ, όπως ξέρετε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την υποδειγματική συνεργασία. Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι το σχέδιο εκτές πηγαίνει σε μια καλή κατεύθυνση, αν και βέβαια έχουμε κάποιες διαφορές σε κάποιες πτυχές. Πρώτα απ' όλα, σημαντικό είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν αμφισβητεί τα υποχρεωτικά στοιχεία της έκθεσης. Ε, θεωρούμε λοιπόν πως θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αξιολόγηση. Μετά από χρόνια εθελοντικής ε, συνεργασίας θεωρούμε ότι έχει φτάσει η στιγμή η Κομισιόν να πάει ένα βήμα παραπέρα. Θα είναι λοιπόν αναγκαίο να, ξεκαθαρί... να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το πλαίσιο το τι επιτρέπεται και το τι όχι όταν μιλάμε για κλινικές ε, αξιολογήσεις χωρίς να υπάρχει περιττή αλληλεπικάλυψη. Κύριε Πρόεδρε, επίσης αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες των ε, κρατών μελών, ειδικά όσον αφορά την ποιότητα και τις ε, κοινέ κλινικές αξιολογήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ομοιόμορφο πεδίο ανταγωνισμού, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει από την μία μέρα στην άλλη. Αυτά τα έχει πει οπωσδήποτε η συγκήτρια, αλλά μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Επίσης η μεθοδολογία της ε, επιστημονικής ε, αποδείξεως θα πρέπει να ε, γίνει ακόμα πιο λεπτομερής. Ειδικά όσον αφορά τα φάρμακα χρειάζεται ένας βαθμός ευελιξίας στο απαιτούμενο επίπεδο αποδείξεως γιατί δεν είναι παντού το ίδιο επίπεδο αποδείξεων διαθέσιμο και θα υποβάλουμε τις σχετικές τροπολογίες και δεν συμφωνούμε εδώ πέρα πλήρως με την εισηγήτρια και αντιλαμβάνομαι πως πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τον κρατών μελών και είναι σαφές ε, πως ε, η προσθέμενη αξία των φαρμάκων εξαρτάται πάρα πολύ από τους οργανισμούς ε, των κρατών μελών. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο εθελοντική συνεργασία στην κλινική αξιολόγηση των φαρμάκων αυτών. Μετά από λίγα χρόνια νομίζω πως μπορούμε να προχωρήσουμε στην ε, υποχρεωτική συνεργασία. Επίσης η περισσότερη συνεργασία και η ψηφιοποίηση είναι κάτι το θετικό, είναι κάτι το οποίο ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια και θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή προδιαγραφή για την ανταλλαγή των ηλεκτρονικών φακέλων των ασθενών ε, έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να έχουν λόγο μόνο οι ειδικοί και όχι οι ίδιοι οι ασθενείς για τα δεδομένα τους τα οποία κυκλοφορούν. Και τέλος, τέλος, κύριε Πρόεδρε, προέκυψε από την ε, καθηγήτρια Άνια Έρκο Κλέρερα από το Πανεπιστήμιο του Ροτερντάμου ότι κάποια φάρμακα είναι πέντε φορές ακριβότερα από άλλα και πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα και στην ε, φαρμακοβιομηχανία και άλλου. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό αυτό για εμάς και θα υποβάλουμε τις σχετικές ε, τροπολογίες γιατί το θέμα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τους ασθενείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παραμείνετε εντός χρόνου. Ο κύριος Πιέχα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Γνωρίζω ότι το θέμα αυτό είναι μια κορυφαία προτεραιότητα υπάρχουν διαφορές γνωμοδοτήσεις και για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως και διαφορετικές απόψεις. Η πρόταση είναι επιμαχή, ειδικά τώρα που το Κοινοβούλιο προετοιμάζει την δική του έκθεση και υποβάλλει τροπολογίες. Θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουμε την συνεργασία μέσω κοινών δοκιμών και κοινών αρχών όταν μιλάμε για κλινικές δοκιμές. Όμως, ο κανονισμός αυτός δεν αφορά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατών μελών και δεν αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Αυτά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όταν δημοσίευσε η Κομισιόν την έκθεση ακούσαμε μόνο τα θετικά αποτελέσματα, περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερος ρόλος για τις οργανώσεις των ασθενών. Όμως, ως Ευρωβουλευτής, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά τα θετικά, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες πτυχές. Το πρώτο τέτοιο ζήτημα είναι το άρθρο 5, το οποίο μιλάει για τη συμπερίληψη ιατρικών συσκευών υψηλότερου ρίσκου. Η αξιολόγηση των συσκευών είναι πολύ διαφορετική από την αξιολόγηση των ιατρικών προϊόντων. Είναι τελείως διαφορετικές. Όμως οι ιατρικές συσκευές ε, κυρίως ε, τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μια λυσίδα προϊόντων, φαρμάκων δηλαδή. Οπότε έχω κάποιες επιφυλάξεις όταν μιλάμε για την συμπερίληψη ιατρικών συσκευών και κάποιες από αυτές απαιτούν ειδική εκπαίδευση για τον χειριστή. Όμως αυτό δεν αναφέρθηκε στην πρόταση. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ιατρικές διαδικασίες δεν μπορούν να τυποποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Επίσης, να επιστήσω την προσοχή σας το ότι έχουμε κάποιους περιορισμούς που εμφανίστηκαν στην τροπολογία 56 Παραδείγματο χάρη, όταν λέμε ότι περιορίζουμε την σύνθεση του πάνελ που θα αξιολογεί. Πρέπει να θυμόμαστε αυτούς που δημιουργούν και αναπτύσσουν τη φαρμακευτική βιομηχανία δηλαδή και επίσης ε, την βιομηχανία ιατρικών συσκευών. Δεν μπορούμε να τους παραλείψουμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε τους στόχους εάν εναρμονίσουμε υπερβολικά ειδικά όσον αφορά την το HDA και τις ιατρικές συσκευές θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην δημιουργήσουμε περισσότερα εμπόδια. Σας ευχαριστώ κύριε Μάισνερ. zunächst ganz herzlich bei der Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα και θα πρέπει να συνεχίσουμε τι εργασίε μα σε αυτό. Θα ήθελα να πω ότι η πολιτική μα ομάδα υποστηρίζει αυτή την πρόταση, να υπάρχει δηλαδή μία ενιαία αξιολόγηση τεχνολογία ε, και όχι ε, 28 διαφορετικέ, 27 στο μέλλον. Ε, ειδικότερα ε, μπορούν να υπάρχουν περισσότερες αξιολογήσεις σε ένα κράτος μέλος, οπότε μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος ε, ο αριθμός. Άρα λοιπόν με ένα κοινό σύστημα έχουμε λιγότερα εμπόδια και κάτι τέτοιο αποβαίνει προς όφελος των καταναλωτών. Ωστόσο τα προβλήματα βέβαια θα τα βρούμε στις λεπτομέρειες και το αντιλαμβάνονται όσοι ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει πολύ ε, σκεπτική στάση από την πλευρά ορισμένων ε, κρατομελών. Για παράδειγμα, η ε, Γερμανία έχει ζητήσει να γίνει μια εξέταση σε ό,τι αφορά την το σεβασμό της αρχής της επικορικότητας. Οπότε ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τη συνεργασία και να μην ε, μπλοκάρει ουσιαστικά μια συμφωνία των Συμβουλίων. Ε, τώρα θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση προ τα ποιο μορφή θα λαμβάνει αυτή η ε, αξιολόγηση. θεωρούμε πως η Επιτροπή δεν έθεσε την δεν εστίασε εκεί που θα έπρεπε. Δηλαδή θα έπρεπε να μας δώσει μια λεπτομερή παρουσίαση του πώ ακριβώς θα υποβάλλονται τα σχετικά δεδομένα ε, για αυτές τις μελέτε. Ε, και νομίζω πως η συγκίτρια τη εκθεσή μας κάνει καλές προτάσεις διόρθωση τη πρόταση τη Επιτροπής. Σίγουρα λοιπόν ε, κινείται προ σωστή κατεύθυνση παρότι υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα. Πάντως, παρότι Υπάρχει με πολύ σκεπτική στάση από την πλευρά ε, των ε, κρατών μελών, δεν θα πρέπει να κάνουμε μια ε, συγκεκριμένη πρόταση ό,τι αφορά να κατανομή των αρμοδιοτήτων συγγνώμη, στο Συμβούλιο, γιατί έχουν ένα είδο αλλεργία εντό εισαγωγικών τα κράτη-μέλη απέναντι σε κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη γενικότερη συμπερίληψη των προϊόντων σε αυτή την αξιολόγηση και των ιατροτεχνολογικών ε, προϊόντων ειδικότερα, ε, θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Γκροστέτ. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα ιατροτεχνολογικά ε, προϊόντα και δεν θα μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε απλώ και μόνο σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα. Υπάρχουν δηλαδή και ζητήματα ω προ την κατάρτιση του χειρούργου, του ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού προσωπικού και ό,τι Και εάν προβλέψουμε υποχρεωτική συμπερίληψη και των ιατροδρομικών ε, προϊόντων ε, στο σύστημα των ε, αξιολογήσεων, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευφυέ από τη δική μα πλευρά, γιατί δεν θα εγγυηθεί οπωσδήποτε μια βελτίωση των αξιολογήσεων. Εγώ ήμουν εισηγήτρια σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και γνωρίζω ποια είναι τα, τα όσα προβλέπονται για την ασφάλεια, για την διεξαγωγή των κλινικών μελετών και ό,τι καθεξή. Οπότε α δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο περαιτέρω εφαρμογή αυτού του κανονισμού και α δούμε μετά τι θα γίνει. Άρα λοιπόν ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα κοινό υποχρεωτικό σύστημα, να υπάρχει ένα συντονισμό μεταξύ των κρατομελών. Κάτι τέτοιο είναι προ όφελο και των ασθενών, αλλά θα πρέπει να δούμε ε, και πού θα αναλάβουν και ποιε αρμοδιότητε τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να επιτύχουν μια γενικότερη βελτίωση για όλα τα κράτη-μέλη. Και αναμένω με ενδιαφέρον τη συνεργασία μα. Κυρία Ριβαζή, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, να επενθυμίσω κάτι στους συναδέλφους. Δεν είναι επαναστατικό το κείμενο. Να συγχάρω την κυρία Καμπεσόν Λουίς για την έκθεσή της και την εξέλιξή της. Συμφωνούμε με τα συμπεράσματά της. Υπάρχει ήδη συνεργασία σε επίπεδο κρατών μελών. Όχι στην περίπτωση της αδειοδότησης, μιλάμε για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας του φαρμάκου ή ε, της ε, ιατρική συσκευή. Αδειοδότηση είναι Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Εδώ βλέπουμε μια προστιθέμενη αξία του φαρμάκου. Και εγώ είμαι στο πεδίο εφαρμογής είναι πολύ σημαντικό αυτά, να συμπεριλάβουμε αυτές τις ιατρικές συσκευές. Γιατί δεν μιλάμε για την διοδότηση, αυτή γίνεται εκτός. Θέλουμε να δούμε ποια είναι η προστιθέμενη υπηρεσία, η προστιθέμενη αξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται επιστημονικές αξιολογήσεις. Και η επιστημονική αξιολόγηση είναι η σύγκριση του νέου φαρμάκου εν συγκρίση με τα ήδη υπάρχοντα. Και εκεί επισημαίνω ότι επί του παρόντος έχουμε ελάχιστα στοιχεία. Αν αυτό το κείμενο είναι καλό, θα προωθήσει τα εργαστήρια, τα φαρμακευτικά να κάνουν συγκριτικές μελέτες, να δούνε ποια είναι η προστεθέμενη αξία του φαρμάκου. Αυτό που έκανε η ΑΣΕΣ στην Γαλλία και άλλοι φορεί στη Γερμανία. Και θα μπορέσουμε να εναρμονίσουμε τα διάφορα πρωτοκόλλα. Οπότε αυτό θα οδηγήσει σε προστιθέμενη αξία όσον αφορά την επιστημονική αξιολόγηση των φαρμάκων από πλευρά συγκρίσεω. Ποιο είναι το σχέδιο εργασία. Θα αφορά όλα τα φάρμακα και όλε τι ιατρικέ συσκευέ. Ουχή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βασιστούμε στα νέα φάρμακα, κυρίως αυτό που αφορά την καινοτομία. Όσον αφορά τον καρκίνο υπάρχουν φάρμακα καινοτόμα και πρέπει να γίνει η μελέτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, όλα αυτά αντίθετα με αυτά που είπα συνάδελφοι δεν μπορεί να γίνουν παρά μόνο αν υπάρχει μεγάλη ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων και υπάρχουν χάρτες που αφορούν την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα ιατρικά εργαστήρια για να γίνει σωστά η εξολόγηση και χρειάζεται διαφάνεια στη συζήτηση. Είναι το DNA το ευρωπαϊκό, η διαφάνεια, η ανεξαρτησία και οι επιστημονικές αξιολογήσεις για να ξέρουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία του φαρμάκου και της ιατρικής συσκευής. Αν κινηθούμε το τρόπος, πιστεύω πραγματικά ότι κάνει πάρα πολύ καλή εργασία σε αυτό το τομέα η συγγήτριά μας να ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κονέτσινα, είναι η επόμενη. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι στην επόμενη συνάντηση πρέπει να εξετάσουμε και τη μείωση του οικολογικού μας ίχνου. Ίσως να χρησιμοποιούμε λιγότερο τον κλιματισμό. Αυτό ένα σχόλιο στο περιθώριο. Και τώρα μπαίνω στο θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως έλεγα, επανειλημμένα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που οδηγεί σε αξιολόγηση ευρωπαϊκή αυτών των συσκευών είναι αποτέλεσμα των αιτήματων των μας του περσινού μας ε, ψηφίσματος όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απλή καταχώρηση των φαρμάκων και των ιατρικών συσκευών γίνεται βάσει αξιολόγηση τη ασφαλεία του. Δεν εγγυάται όμω ότι τα νέα φάρμακα είναι ένα βήμα προέδρου. Όπω έλεγε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία μάλλον, πρόσφατα τον Μάιο του 2014 οι τεχνολογίες ιατρικές θα πρέπει να οδηγούν σε μεγαλύτερη πρόσβαση στις θεραπείες. Σε διάφορα κάτι μέλη οι αποφάσεις είναι διαφορετικές όσον αφορά τα φάρμακα και ασθενεί για τα ίδια φάρμακα. Οπότε είναι σαν η θέση διάφοροι ασθενεί. και αυτό δημιουργεί και κάποια σύγχυση. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Συνήθω αποφάσεις παίρνουν μικρές ομάδες ατόμων όμως. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στην ε, αξιολόγηση αυτών. Θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμό των πόρων και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και θα έχουμε καλύτερη αξιολόγηση που θα είναι αποτελεσματικότερη ε, για όλα τα κράτη-μέλη και θα απεφευθούν αλληλεπικαλύψει και τα μικρά κράτη-μέλη βοηθηθούν έτσι όπω το δικό μου που δεν έχουν επαρκή πόρου και αρμοδιότητα για να κάνουν πολύ ποιοτική αξιολόγηση. Δέχομαι θετικά την πρόταση τη ηγήτρια. Εδώ και ένα χρόνο συνεργαστήκα μαζί τη όσον αφορά την την πρόσβαση στα φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μ' αρέσουν οι βελτιώσει που έχουν γίνει όσον αφορά την ταυτοποίηση τη προστιθέμενη αξία των φαρμάκων τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, θα πρέπει οι ασθενεί να μπορούν να συμμετέχουν στην όλη διακυβέρνηση και να σκεφτούμε και τι σπάνιε ασθένειε όσον αφορά τα φάρμακα. Επί καιρό ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να επεξεργαστούν τη δυνατότητα αξιολόγηση των διαφόρων τεχνολογιών που ήδη έχουν δημοσιευτεί. Η παρούσα πρόταση εδράζεται επί μια αξιολογήσεω ή αποφάσεω χωρί δυνατότητα βελτίωση. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό κάτι. Έχω απογοητευτεί επί κάποιων σημείων στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γίνεται λόγο για μια υποχρεωτική αξιολόγηση των ιατρικών συσκευών και των φαρμάκων. Δεν άλλαξαν τα πράγματα σε αυτό το μέτωπο. Ε, προσβλέπω σε συνέχιση συνεργασία με την συγγήτρια. Δεν θα είναι απλά τα πράγματα, αλλά πρέπει να πείσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο ώστε να συμμετάσχουν στην προσπάθεια και θα πρέπει να καταλάβουμε σαφώ περί τίνο πρόκειται η αρχική πρόταση. Συμφωνώ μαζί σα πλήρω, λέει ο Πρόεδρο, για την οικολογική προσέγγιση που είπατε, για το κλιματισμό. Να εγκαταλείψουμε, όπω έκανε και ο Ντέμε Μάκερ, και τι πλαστικέ φιάλε ύδατο και να φέρουμε τι δικέ μα φιάλε. Ο κ. Πεντιτσίν είναι επόμενο που έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή τη και την εισηγήτρια ευχαριστώ για τη δουλειά που έκανα μέχρι τώρα, που κατά την άποψή μα είναι πολύ καλή. Η εισηγήτρια κ. Καμπεζόν αναφέρθηκε στην ανεξαρτησία των αξιολογήσεων. Συμφωνούμε με αυτήν. Πιστεύουμε εξάλλου ότι η εθελοντική συνεργασία που μέχρι τώρα χαρακτήρισε τις προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών μελών σε αυτό το πεδίο. Ήταν θεμελιώδη σημασία για να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο. όμω, τώρα είναι και η ώρα να επισημοποιηθεί το πλαίσιο δράσεω, να κάνουμε ποιοτικό άλμα ε, προ τον υποχρεωτικό χαρακτήρα και να μιλήσουμε για επέκταση του πεδίου εφαρμογή ίσω για τι ιατρικέ συσκευέ, medical devices. Με έκπληξη άκουσα αυτά που είπε ο συνάδελφο Πιέκα του ECR που αναφέρθηκε σε υπερβολική εναρμόνιση Πάλι καλά που ήμασταν εμείς οι αντιευρωπαϊστές. Είναι σημαντικά αυτά. Πρέπει όλοι να τα μοιραζόμαστε. Οι μόνοι που, τους συναδέλφους που κατάλαβαν πραγματικά περί τίνο συζητάμε είναι οι συνάδελφος Ριβαζή και Κονέτσνα. Διότι εδώ δεν μιλάμε για διοδότηση. Προτείνω λοιπόν στους συναδέλφους του ECR και του ΕΛΚ και της ΑΛΔΕ να εμβαθύνουν λίγο καλύτερα στο θέμα και να δώσουν καλύτερα επιχειρήματα σε αυτά που λένε. Εμείς είμαστε υπέρ της προτάσεως διότι αντιστοιχεί σε δύο ουσιαστικές ανάγκες. Αυτή για τη μείωση των δαπανών και της πατάλης και εξορθολογισμό των πόρων από την άλλη. Τα δύο πράγματα δημιουργούν, έχουν αποτέλεσμα πιο ευέλικτες διαδικασίες και καλύτερες δυνατότητες θεραπείας για τους ασθενείς. Ταυτόχρονα υπενθυμίζω ότι το ιταλικό πείραμα που ήταν κάτι θετικό. Πολλές περιφέρειες Ιταλίας ήδη δημιούργησαμε κάποια διαδρομή όπως το Βένετο, η Λομβαρδία, η Τοσκάνη και το Λάτσιο και στα νότια στην Πούλια. Ε, χρειάστηκε όμως ένα συντονισμό εθνικός. Αν όλα αυτά τα ανεβάσουμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ανάγκη συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ιταλία έχει πολλά να δώσει σε αυτό. Την εμπειρία που έχει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ερευνητικών προγραμμάτων. Δεν πιστεύω ότι έχει καλυφθεί επαρκώς από την παρούσα πρόταση. Θα εργαστούμε από αυτού και ελπίζουμε το ταχύτερο δυνατό να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, η κυρία Μιλά, τελευταία σκιώδηση συγκεκριά. Madame Mélin. Κυρία Μιλέν δεν βρίσκεται εντός αιθούσης. Τα μέλη της Επιτροπής σε δίλεπτο. Η κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ. Ε, ομιλώ εκ μέρους του συναδέλφου Πεταλίζα γιατί βρίσκεται σε μια ε, συνεδρίαση ε, στο Μοναχό, οπότε διαβάζω τα όσα μας ε, υποστηρίζει την πρόταση ε, της Επιτροπής ε, και θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιμο το τμήμα εκείνο το οποίο θέλει ένα καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ ΕΜΕΣ και ε, των οργανώσεων που προβαίνουν στι αξιολογήσει. Γιατί κάτι τέτοιο θα μπορέσει να επιφέρει πραγματικά θεραπευτικέ βελτιώσει και για του ασθενεί. Ωστόσο, ο κύριος Πέτερ Ελίζε θεωρεί ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, ε, το επίπεδο των σχετικών υπηρεσιών είναι ε, διαφορετικό στα διαφορετικά κράτη-μέλη, οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία συγκριτική θεραπεία. Και εάν υπάρχει αντίρρηση σε ό,τι αφορά αυτήν τη μία αναλλακτική θεραπεία, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν το υψηλότερο πρότυπο που προβλέπουν τα ίδια. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ένα αιτιολογημένο opt-out, δηλαδή η δυνατότητα να μη συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα. Ε, για νομικούς, νομοθετικούς λόγους δεν θα πρέπει να το ενισχύσουμε το opt-out, αλλά θα πρέπει να παραμείνει ως δυνατότητα. Μετά στην ε, πρότασή της Επιτροπή αναφέρει ότι η σχετική ε, αρμόδια Επιτροπή θα αποφασίζει είτε με πλειοψηφία είτε ομόφωνα. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό περαιτέρω όμως, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε αν θα είναι απόλυτη πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία, αφού υπάρχει ιδιαίτερη αντίρρηση από την πλευρά των κρατών μελών. Κατά δική μας άποψη, ακριβώς για αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να υπάρχει να ισχύει πλειοψηφία, ομοφων... Ε, πλειοψηφία δύο τρίτων ή ομοφωνία, αλλά ειδική πλειοψηφία. Ε, από εκεί και μετά θα πρέπει να υπάρχει ε, η δυνατότητα ακύρωσης, ε, προβλέπει η πρόταση η δυνατότητα ακύρωση από την πλευρά της Επιτροπής, η οποία έχει ληφθεί ακόμα και ομοφόνο από τη σχετική αρμόδια Επιτροπή. Θεωρούμε πω κάτι τέτοιο είναι δυσανάλογο. Δηλαδή, εάν έχει ληφθεί μια απόφαση από την αρμόδια Επιτροπή ε, με ειδική πλειοψηφία, τότε μόνο υπό εξαιρετικέ περιστάσει θα είναι δυνατόν να αμφισβητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εκεί και μετά, και τελευταίο σημείο, ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Γιατί ο κύριο Επετελίζε θεωρεί ε, πω η πρόταση τη ε, Επιτροπή αλλά και η πρόταση του εισηγητή δεν είναι ιδανικέ. Εδώ πρόκειται για μια διαδικασία η οποία προβλέπει δηλαδή έλεγχο, αλλά σε ό,τι αφορά τι πτυχέ ασφαλεία. Και ούτω μια τέτοια αξιολόγηση σε ό,τι αφορά τι πτυχέ ασφαλεία δεν μπορεί να ισοδυναμεί με μια αξιολόγηση ε, τεχνολογιών υγείας και γι' αυτό ενδεχομένως θα χρήσιμο θα ήταν να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ε, διαδικασία αξιολόγησης ε, των τεχνολογιών υγείας αφού δημιουργήσουν τις δικές τους αξιολογήσεις στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Καπούτα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το δικαίωμα στην υγεία και στην περίθαλψη είναι κάτι που πρέπει να εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους πολίτες της. Σύμφωνο λοιπόν με την τροποποίηση του κανονισμού και τις προτάσεις της Σολεδάδ νομίζω ότι στην αρχική έκθεση υπάρχει μια συνένεση για καλύτερη πρόσβαση σε φάρμακα και ιατρικά προϊόντα και στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο να βελτιώσουμε την αγορά και να αποφύγουμε της στρεβλώσεις αλλά να αυξηθεί η ποιότητα της καινοτομίας και της τεχνολογίας να ορίσουμε προτεραιότητες στην έρευνα και πρόσβαση στα προϊόντα αυτά. Είμαι υπέρ της ε, ανάπτυξης ε, των ιατρικών τεχνολογιών και της αξιολόγησής τους και βεβαίως ε, μια συνεργασία δεσμευτικής φύσης και η εγγύηση υψηλή ποιότητας αξιολόγησης βεβαίω πρέπει να είναι ανεξάρτητη και με διαφάνεια. Η Κομισιόν θα είναι υπέρ τη σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και της χρηματοδότηση που πρέπει να είναι δημόσια και ανεξάρτητη αλλά δεδομένου του ότι τα φάρμακα είναι πολύ ευαίσθητο τομέα. χρειάζομαι Χρειάζεται περαιτέρω προφύλαξη για να μην αποφεύγει ο κόσμος τις υποχρεώσεις του. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην Κομισιόν, κυρία Άμπελα. Έχει τον λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και σας ευχαριστώ για την γενική σας στήριξη για την συνεχιζόμενη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα αυτά και για την ίδια την πρόταση και να σας υπενθυμίσω ότι η πρόταση αυτή βεβαίως ε, ανταποκρίνεται σε έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν βεβαίως δεν ξεκινάμε από το μηδέν, έχουμε πάνω από 20 χρόνια συνεργασίας στην ε, αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας ε, και γι' αυτό ακριβώς τώρα πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Και συμφωνούμε με τις απόψεις του εισηγητή ότι η πρόταση αυτή αφορά την αύξηση του επίπεδου επιστημονικών στοιχείων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα ιδιαίτερα να σχολιάσω κάποια συγκεκριμένα σημεία που ακούστηκαν και θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα του πεδίου της εφαρμογής. Γιατί οι απόψεις ε, δίστανται. Από την πλευρά της Κομισιόν προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στα προϊόντα τα οποία θεωρούσαμε ότι έχουν τη μεγαλύτερη προσθέμενη αξία, διασυνοριακές πτυχές και να υπάρχει και μια νομική βεβαιότητα. Γι' αυτό ασχοληθήκαμε και εστιάσαμε στα κεντρικώς αδειοδοτούμενα ιατρικά προϊόντα και τις ιατρικές συσκευές υψηλού κινδύνου. Καθορίσαμε προσεκτικά το πεδίο, ακούγοντας τους διάφορους ενδιαφερόμενους, ε, τις ανησυχίες ε, του κλάδου. Θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή είναι αναλογική. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω κάποιους ομιλητές ότι όσον αφορά τις ε, διαφορετικές πόριες ε, προς την αγορά. Το λάβαμε υπόψη αυτό στις ιατρικές συσκευές. Γι' αυτό είναι πιο περιορισμένο το πεδίο και δεν παρεμβαίνουμε με τον σχετικό κανονισμό όσον αφορά τον χρόνο. Θα ήθελα να πω επίσης λίγα λόγια ε, για τα υποχρεωτικά στοιχεία αυτής της πρότασης γιατί είναι κάτι το σημαντικό. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ποιος είναι ο βασικός στόχος της πρότασής μας. Θέλουμε ακριβώς οι καλύτεροι ειδικοί να συνεργαστούν και το σκεπτικό είναι η δουλειά αυτή να χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο και να μην επαναλάβουμε δουλειά που έχει ήδη γίνει. νομίζω ότι είναι σημαντικό στο πλαίσιο αυτό να ξεκαθαρίσουμε το τι εννοούμε με την κοινή έκθεση κλινικής αξιολόγησης. Μία έκθεση δηλαδή γενικής φύσεως δεν πρόβλημα. να πούμε ότι θα λέμε ότι μία τεχνολογία είναι καλύτερη από άλλη, αλλά μία έκθεση πιο γενική και θα ήθελα να σχολιάσω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Λίζα για τις συγκρίσεις. Θα είναι απολύτως δυνατόν να κοιτάξουμε διαφορετικά συγκριτικά στοιχεία εντός της έκθεσης. Από την άλλη, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τα κράτη-μέλη όταν ενσωματώσουν ε, στο εθνικό του σύστημα την δουλειά αυτή για να δουν και τα μη κλινικά στοιχεία, να δουν τη γενικότερη αξιολόγηση των συμπερασμάτων στην εθνική τους διαδικασία. Και νομίζω ότι συμφώνησαν ε, οι βουλευτές ότι δεν ε, επηρεάζεται εδώ πέρα η αρμοδιότητα των κρατών μελών για την υγεία, την τιμολόγηση και την καταβολή των εξόδων. Θα ήθελα κατόπιν να σταθώ στον ρόλο της Κομισιόν γιατί ακούστηκαν και κάποια σχετικά ερωτήματα. Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι σύμφωνα με την πρόταση, αυτό το οποίο περιμένουμε εμείς είναι τα κράτη-μέλη να κάνουν την τεχνική δουλειά. Οι ειδικοί στα κράτη-μέλη θα κάνουν τεχνική δουλειά. Η Κομισιόν θα απλά θα κοιτάει ότι ε, ακολουθείται σωστά η διαδικασία και θα δημοσιεύσει την έκθεση μόλις ολοκληρωθεί. Και έτσι έρχομαι στο θέμα της ισορροπίας μεταξύ της βασικής νομοθεσίας και των εφαρμοστικών κανονισμών στα κράτη-μέλη. Και βέβαια έχουμε τα βασικά στοιχεία τα οποία θα συμπληρωθούν με κάποιες πράξεις κατά εφαρμογή και κατά εξοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό πράγματι να υπάρχει η σωστή γνωμοσύνη όταν αναπτύσσουμε την δευτερογενή νομοθεσία. Γι' αυτό ακριβώς βασιζόμαστε στη δουλειά που γίνεται στην κοινή δράση UNETA. Γι' αυτό βασιζόμαστε στην πύρα των εθνικών αρχών. Να σας διαβεβαιώσω πως ε, η διαφάνεια είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειά τη ε, Κομισιόν και αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Όσον αφορά την ψηφοφορία, διαπιστώνουμε ότι έχει υπάρξει πρόταση να αυξηθούν τα κατόφλια. Εμείς θα θέλαμε μια συνενετική διαδικασία και αυτό νομίζω σχετίζεται με αυτό το οποίο είπα για την φύση και το πεδίο εφαρμογή ε, των εκθέσεων. Πρόκειται για μια γενική έκθεση που ελαμβάνει τα πάντα, οπότε θα θέλαμε να υπάρχει συνένεση στην ομάδα συντονισμού. Ποιος θα κάνει τη δουλειά. Κοιτάξτε, όταν μπει σε ένα νομικό πλαίσιο πρέπει να υπάρχει λογοδοσία και απαραίτητη ευθύνη. Γι' αυτό επιλέξαμε την λύση οι αρμόδιες εθνικές αρχές να είναι μέλη της ομάδας συντονισμού και έτσι θα έχουμε τους καλύτερους ειδικού για να κάνουν την τεχνική δουλειά. Αυτό λέει η πρότασή μας και νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τα όσα θα θέλαμε δηλαδή την βέλτιστη χρήση των πόρων. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα ξανά στην κυρία Καμπεθόν Ρουής. Θα είμαι πάρα πολύ επιγραμματική. Ευχαριστώ όλου του και ηγητέ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικοδομητική του στάση που θα μα επιτρέψει να πετύχουμε την αναγκαία συμφωνία ε, επί τη βάση του γεγονότος ότι όλοι έχουμε κάτι σχετικό μας απασχολεί είναι έξοχη βάση αυτή για τις εργασίες μας. Να, δεν θα πρέπει να ρισμονούμε ότι πρόκειται περί επιστημονικής εργασίας ε, υψής της ποιότητας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη για όλους, για τη βιομηχανία που μπορεί να κερδίσει και αυτή διότι θα υπάρχει ένα είδος πιστοποίησης που θα οδηγεί σε προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Και μετά θα έχουμε μια βελτίωση για τους ασθενείς και την πρόσβαση που θα έχουν στην τεχνολογία αυτή. Αυτό είναι ο πυρήνας της ε, επιστημονικής προσπάθειας να καταβληθεί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι οι επιστήμονες και όλα αυτά αυτή η προσπάθεια θα καταλήξει σε κάτι υποφελές για όλους. Ευχαριστώ. Οπότε ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Η υποβολή τροπολογίων είναι 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 13 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο και Ψηφοφορία στην Ολομέλεια αναμένεται 1η Οκτωβρίου. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτό το σημείο και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επόμενο σημείο, ανάπτυξη υποδομίων, ε, διαφόρων υποδομών, ε, ώρα για δράση. Θα δώσουμε το λόγο στον Κρίστιαν Καλεμόζο, στην Κρίστιαν Καλεμόζο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω ε, να είμαι ε, πικοδομητική. Όσο αφορά τα αναλλακτικά καύσιμα, είχαμε μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Τρανς. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πρέπει να τονίσουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Να έχουμε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα στη Συμφωνία των Παρισίων έχουμε υποχρεώσει την Ευρώπη να μειώσει τα αέρια του θερμοκηπίου και τις εκπομπές σχετικές κατά 20% μέχρι το 2020 και 40% μέχρι το 2030. Για να το πετύχουμε αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε εναλλακτικέ ε, πηγές, εναλλακτικά καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται και για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε μια εύρυθμα λειτουργούσα υποδομή και αυτό συζητούμε εδώ ε, να τονίσω ότι καλωσορίζω το σχέδιο δράσεως αυτό για, για τα ανακτικά κάψιμα. Είναι προϋπόθεση να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές στην Ευρώπη. Για κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε φιλόδοξη προσέγγιση να αφορά τα εθνικά σχέδια. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλέ διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Πάνω απ' όλα αυτό είναι ευθύνη των κρατών μελών όμως. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν, θα πρέπει να εφαρμόσουν τους στόχους που έχουμε θέσει. Θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη γι' αυτό. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων των κρατών μελών. Δεν ανταποκρίνονται όλες οι χώρες στις υποχρεώσεις τους και θα είναι κρίσιμο κάτι τέτοιο αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Χρειαζόμαστε συντονισμένη προσέγγιση ε, Λοιπόν, είναι έτοιμος για τα εναλλακτικά καύσιμα ο κόσμος, η βιομηχανία είναι έτοιμη, έχει τεχνικές λύσεις, αλλά περιμένουν να έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν. Αυτό είναι το αστείο. Όλα εξαρτώνται τώρα από τα κράτη-μέλη ε, που πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές, ούτω ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ωφεληθούν θέλουμε να έχουμε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Αν θέλουμε να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εναλλακτικά κάψιμα που είναι στη διάθεσή μα. Αυτό που κάνω λοιπόν στο σχέδιο γνωμοδοτήσεώ μου για την Επιτροπή Μεταφορών είναι να καθιστώ σαφέ ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε τώρα, θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Έτσι παροτρύνω τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν και να εφαρμόσουν να υλοποιήσουν τις υποδομές για τα αναλλακτικά καύσιμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε ε, πάρα πολύ ε, τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης, πολύ ταχεία φόρτιση στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και δεν κάνουν αρκετά τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να τονίσουμε λοιπόν στη γνωμοδότησή μας ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούν τα κράτη-μέλη και πρέπει να γίνει αυτό, διότι πρέπει να μπορεί να ξεκινήσουν και οι καταναλωτέ και οι επιχειρήσεις. Δεν θα πω πολλά περισσότερα. Πιστεύω ότι είναι όλα πάρα πολύ ξεκάθαρα. Θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Θα πρέπει να κινηθούμε τάχιστα και θα πρέπει επίσης να δραστηριοποιηθούν και τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν υποσχεθεί ότι θα το κάνουν αυτό. Υποσχέθηκαν, αλλά τώρα πρέπει να το υλοποιήσουν. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εμείς εστιαζόμαστε επί της εξασφαλίσεως του ότι θα κινηθούμε κατάλληλα λαμβάνοντας υπόψη πτυχές περιβάλλοντος και κλίματος. Βέβαια υπάρχει και δυνατότητα βιομηχανική για τα κράτη-μέλη. Πρέπει να τονιστεί. Ελπίζω να υποστηρίξετε την γνωμοδότησή μου. Εγώ ίδια ε, κάνω κάποιες συστάσεις, έχω κάποιες τροπολογίες, δεν πάω συμπεριλάβω τα πάντα. Ε, περιμένω να δω ποιες είναι οι δικές σας συνεισφορές, τις περιμένω και ελπίζω να μπορέσουμε να είμαστε φιλόδοξοι και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξεκινήσουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να ασκήσουμε κάποιες πιέσεις επ' αυτόν, ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει ε, στη Συμφωνία των Παρισίων. Για τους συγητές έχουμε λοιπόν τρία λεπτά, για τις άλλες συνεισφορές δύο λεπτά. Ασκιώδη συγητής τώρα, ο πρώτος, αντί του κυρίου Γκριμπ, η κυρία Ζώμα έχει το λόγο που εκπροσωπεί το Ευχαριστώ Πρόεδρε. αγαπητοί συνάδελφοι, προσωπώ εδώ τον συνάδελφο Δήπο, ο οποίος ε, μου διαβίβασε το κείμενό του στα αγγλικά, αφού δεν μιλάω πολωνικά. Άρα λοιπόν, ε, συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε την οδηγία σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά κάψιμα και την υποδομή του το 2014 και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφθορτικά προβλήματα στο επίπεδο της εφαρμογής της. Υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις ενώπιον μας ε, και το κυριότερο είναι η έλλειψη ε, παρκούς και αξιόπιστης υποδομής για αυτά τα καύσιμα. Ωστόσο, η οδηγία δεν εστιάζει μόνο ε, στην υποδομή φόρτισης, αλλά και σε άλλα εναλλακτικά καύσιμα. Ε, αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο, θα είναι ε, σημαντικά για την μείωση ε, της ε, μόλις από τα, των εκπομπών καυσίμων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές μεγάλης απόστασης. Επίσης, θα πρέπει να προωθεί περισσότερο το LNG στους διευρωπαϊκούς διαδρόμους. Θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη λοιπόν υποδομή και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατά συνόπια θα πρέπει να υπάρξει συμπερίληψη αυτής της πτυχή στο μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται αυτέ τι προτεραιότητε και στου προπολογισμού και ε, στου στόχου των θεσμικών οργάνων. Επίση, θα πρέπει να εστιάσουμε και να προωθήσουμε συνέργειε. Ε, και ε, ας ε, μην ξεχνούμε ότι αυτή την περίοδο η, ε, η Επιτροπή προετοιμάζει μια πρόταση σε ό,τι αφορά τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, οπότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι δύο προτάσεις, η παρούσα και εκείνη για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, θα πρέπει να είναι ε, συντονισμένε μεταξύ τους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Δερσμακέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά την ε, κυρία Μόζερ, την εισηγήτρια για αυτή την έκθεση. Όπως ε, λέει και η Επιτροπή, αλλά όπως διαπιστώνουμε και εμείς, ε, ορισμένα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν περισσότερες προσπάθειες εάν θέλουμε να, έχουμε, να επιτύχουμε κάποια στιγμή το στόχο της ε, κινητικότητας χαμηλών ή ακόμα και μηδενικών εκπομπών. Συμφωνώ με αυτόν τον στόχο και συμφωνώ με το ότι θα πρέπει να γίνει μια αναπροσαρμογή των αποδομών μας. Αυτό είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε τους ε, κλιματικούς μας στόχους αλλά και προκειμένου να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ε, στο διεθνέ περιβάλλον. Εάν θέλουμε δηλαδή να έχουμε εδώ σημαντικό ρόλο στην αυτοκινητοβιομηχανία ανά τον κόσμο, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η ζήτηση για τέτοιου είδους οχήματα θα αυξηθεί. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η δική μας τεχνολογία να παραμείνει επίκαιρη. Η συγγήτρια αναφέρει ότι ε, κυρίως η φόρτιση αυτών των οχημάτων γίνεται είτε συνεργασία είτε ε, στο σπίτι. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες δυνατότητες εφόρτισης ε, και μάλιστα κατά μήκο ε, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν οχήματα χαμηλών μηδενικών εκπομπών, τα οποία θα παραμένουν χαμηλών μηδενικών εκπομπών στο σύνολο του κύκλου ε, ζωής τους. Ε, υπό αυτές τις προϋποθέσεις μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια πρόταση. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ ε, και στο ζήτημα της ενεργειακής ουδετερότητας. Ε, δηλαδή, πρωτού προβούμε στην πλήρη μετάβαση στην ενεργειακή ουδετερότητα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή η μετάβαση θα διαρκέσει λίγο χρόνο. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε και λίγο ποιε είναι οι εναλλακτικέ χαμηλών εκπομπών για, την, για το ενδιάμεσο διάστημα. Και α μην ξεχνούμε εδώ ότι υπάρχουν και δημικέ κοινότητε αλλά και κράτη-μέλη ε, για τα οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο πλαίσιο ε, και ιδιόρυθμο δηλαδή. Εγώ στην ε, Φλάνδρα, από την οποία κατάγομαι, διαμένω σε μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλά πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα, σε σύγκριση για παράδειγμα με τη Σκοτία ή αλλού. Οπότε και αυτή η πτυχή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους ε, στόχους ε, που θέλουμε να θέσουμε σε ό,τι αφορά την ε, πώληση των σχετικών ηλεκτροκινητών οχημάτων. Αφού λοιπόν ο στόχος μας είναι να αυξηθούν οι σχετικές πωλήσει, θα πρέπει να δημιουργήσουμε την κατάλληλη υποδομή, αλλά όλα τα υπόλοιπα που ρυθμίζουν τους νόμους της αγοράς και της ζήτησης δεν θα πρέπει να τα επηρεάξουμε, θα πρέπει να τα αφήσουμε στην αγορά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος είναι ο επόμενος σχέδιος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω κάποια λόγια. Κατά το παρελθόν, το 2013, όταν διαπραγματευτήκαμε την οδηγία αυτή για τις υποδομές, για τα εναλλακτικά κάψιμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει στόχους υποχρεωτικούς στόχους και που θα έπρεπε να επιτευχθούν μέχρι το 2020. Δυστυχώς έγιναν κάποιοι συμβιβασμοί εν μεταξύ όταν συζητούσαμε αυτά στο Συμβούλιο. Θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε τους συμβιβασμούς αν οι στόχοι μετα... κάποιοι στόχοι μπορούν να μετακινηθούν για το 2025. Για άλλους δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για τους υποχρεωτικούς στόχους. Στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε κάποιες προθεσμίες για στρατηγικές εθνικές που μπορούν να δημιουργηθούν στα πλαίσια αυτά. Δυόμιση χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει αυτό. Το συζητήσαμε το θέμα στο Κοινοβούλιο το 2016, το 2017 τα αποτελάσματα είναι αξιοθρύνητα. Δύο κράτη-μέλη δεν έχουν καν στείλει εθνικές στατικικές. Μεταξύ άλλων κρατών μελών, μόνο οκτώ έχουν θέσει κάποια εθνικά πλαίσια πολιτικών για το ζήτημα αυτό. Και δεν καλύπτουν όλη την επικράτειά τους. Τώρα, εάν πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό δεν έχουμε πετύχει τους τεθέντες στόχους στον τομέα των μεταφορών. Αν δούμε σε ποιο βαθμό εξαρτώμεθα ακόμα από τα ορυκτά κάψιμα και τα κάψιμα από τα απορριχτές πηγές θα πρέπει να δούμε ότι χρειαζόμαστε ένα πλήρες δίκτυο, ολοκληρωμένο, comprehensive network, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν γνωρίζουμε ότι οι στόχοι για τα αναλλακτικά καύσιμα είχαν προβλεφθεί τελικά να επιτευχθούν το 2025, εάν συνεχίσουμε αυτούς τους ρυθμούς δεν θα πετύχουμε κανέναν από αυτούς τους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει διασυνδεθεί, δεν θα έχουμε τα αναλλακτικά καύσιμα, θα εξαρτόμεθα από από τα ορυκτά καύσιμα και όλα αυτά διότι τα κράτη-μέλη δεν είναι ικανά να πετύχουν τους στόχους στον τομέα αυτό ούτε τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Δέκα κράτη-μέλη δεν έχουν δείξει την παραμικρή φιλοδοξία για τη δημιουργία υποδομής για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Μιλάμε επίσης και για τα κτίρια, για τα τα που θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας. Μιλάμε εκτενώς για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις μεταφορές στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη τις μεταφορές ε, μέσω ε, των ποταμών. Γι' αυτό προτείνω να κινητοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα TNT στην Ευρώπη. Και γι' αυτό θα πρέπει οι στόχοι που θα τεθούν να είναι υποχρεωτικοί, διότι για την ώρα τα κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει τίποτα μακροπρόθεσμα επί της εθελοντικής βάσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη των υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα που παρουσιάστηκε στο δεύτερο πακέτο για την κινητικότητα σίγουρα ένα σημαντικό έγγραφο που περιγράφει τις απαιτήσει για επενδύσεις, συγκεκριμένες απαιτήσει Συμμεριζόμαστε τις γενικές ε, ανησυχίε που εκφράζονται όσον αφορά την άνοιξη των υποδομών για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Κατά την άποψή μα, πρέπει να είναι ένα απαραίτητο στοιχείο ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου. Δυστυχώ γνωρίζουμε ότι δεν έγινε αυτό πάντα, όπως είδαμε και στην Ιταλία και από άλλα κράτη-μέλη, που μέχρι τώρα, μέχρι τώρα, κυρίως στην Ιταλία ισχύει αυτό, έχουν προωθήσει το φυσικό αέριο. Ε, όσον αφορά τις ε, υποδομές τους για στα πλαίσια της λειτουργικής υποδομής που πρέπει να έχει υλοποιηθεί. Λοιπόν, υπεθύμιζαν και συνάδελφοι, έχουμε ακόμα βασιστεί στα ορυκτά καύσιμα και δεν έχουν εναρμονιστεί οι μεταφορές και στη χώρα μου και όχι μόνο. Τα 95% των συστημάτων μεταφοράς στην Ευρώπη βασίζονται σε συμβατικά ορυκτά καύσιμα. Ο κανονισμό είναι καλή αφετηρία για να συμβάλλουμε σαν Επίτροπη Περιβάλλοντο στην προσπάθεια που γίνεται. Συμφωνώ με την εισηγήτρια. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ευνοήσουμε λύσει για την ευφυή φόρτιση βάσει συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κυρίω ότι πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από αυτό που προβλεπόταν από τι ελάχιστε προδιαγραφέ στα πλαίσια τη παροχή ενέργεια στα κτίρια σύμφωνα με την οδηγία που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων για τα σημεία φόρτισης εστιαστικά κέντρα και που θα είναι πρόσβαση ε, των πολιτών. Πρέπει να το εξασφαλίσουμε αυτό. Ε, ελπίζω να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση όπου η κινητικότητα και οι υπηρεσίε φόρτιση να έχουν εντοπιστεί σαφώ και να είναι ακρογωνία λήθο για, για την κινητικότητα. Χρειάζονται πριν και μετά το 2020 επενδύσει. Κατά την άποψή μου όμω δεν να υπάρχουν, δεν υπάρχουν εμπόδια στο τεχνικό επίπεδο. Ποιο είναι το πραγματικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε, η διαθεσιμότητα η πολύ περιορισμένη των ηλεκτρικών ε, οχημάτων στην αγορά. Περιθωριακέ είναι οι πωλήσει 1% του 2017 για τα νέα αυτοκίνητα και τα κέρδη για το περιβάλλον και τον αέρα που αναπνέμε ε, πόρο απέχουν από τον υλοποιηθούν. Και συγχαίρω τη συνάδελφο Ντάλη που κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά για τον νέο κανονισμό για τα, για τα οχήματα σχετικά και ελπίζω να δώσει μεγαλύτερη υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο γύρος των σκιωδών και τώρα πάμε στις άλλες συνεισφορές από τα μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Ντάλη είναι η πρώτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Σχάλντε Μόσα για τις εξαιρετικές ε, προτάσεις της. Θεωρώ ότι το σχέδιο δράσης ε, της Κομισιόν είναι μια πολύ σημαντική συμπληρωματική πρόταση ε, συμπληρωματική στην αναθεώρηση της πρότασης για το διοξείδιο του άνθρακα από το αυτοκίνητο και βεβαίως πολύ συχνά λέμε πως ένα από τα σοβαρά εμπόδια όσον αφορά τα οχήματα χαμηλών και μηδενικών οικομών είναι οι υποδομές όμως δεν είναι αυτή η συνολική εικόνα. Θα ήθελα να σας παραπέμψω σε μία ανάλυση που έκανε η πλατφόρμα ηλεκτρονικής ε, κινητικότητας που λέει πως είναι χαμηλή η διαθεσιμότητα των οχημάτων ε, αυτών για τις χαμηλές πωλήσει και βρήκε συνολικά πως υπήρχαν πέντε ηλεκτρικά ε, οχήματα Α, με συγχωρείτε υπήρχαν πέντε σημεία φόρτισης ε, για κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον δρόμο αλλά πέντε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με συγχωρείτε ανά σημείο φόρτισης ε, αλλά το θέμα ήταν που βρίσκονταν αυτά και τώρα θα υπάρχουν ε, προσεχώ ε, γύρω στα 10 αυτοκίνητα ανά σημείο φόρτιση. Συμφωνούμε όμως ότι χρειάζονται δημόσιε επενδύσει ε, στι υποδομέ πριν και μετά το 2020 καθώ οι πωλήσει αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών θα αυξηθούν. Εδώ πέρα λοιπόν έχει σημασία ο χρονισμό και η διαλειτουργικότητα και πρέπει να συνεργαστεί η βιομηχανία με τα κράτη και τους δήμους. Και εδώ πέρα θεωρούμε ότι η δουλειά του δημόσιου τομέα είναι να εντείνει τις προσπάθειες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και να κινητοποιήσει τις δημόσιες επενδύσεις, να στείλει τα σωστά κίνητρα και να προωθήσει τις πράσινες δημόσιες επενδύσεις. Υπάρχει και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα που πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει επιχειρηματικό μοντέλο για την εγκατάσταση τέτοιων σταθμών φόρτισης και να αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ. κυρία Μάισνερ. Να ευχαριστώ πάρα πολύ ζήτησα τον ε, λόγο. Νόμιζα ότι ήταν άλλος ο σκιώδης εισηγητής μας ε, που δεν είναι εδώ. Λοιπόν, παρακολούθησα το θέμα αυτό για την Άλντε το 2014 όταν ε, εγκρίθηκε και είμαι και σκιώδης εισηγητή στην Επιτροπή Μεταφορών. Κοιτάξτε, πράγματι η νομοθεσία του 2014 δεν ήταν τόσο φιλόδοξη όσο θα θέλαμε. Η πρόταση της Κομισιόν προέβλεπε μια εφαρμογή νωρίτερα και πιο φιλόδοξη και το Κοινοβούλιο το ίδιο και πραγματικά πάρα πολλά πράγματα στον διάλογο με τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο γιατί εμείς θα θέλαμε βεβαίως ε, να τα αναθεωρήσουμε αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί ακόμα έχουμε τη φάση της εφαρμογής μέχρι το 2020 ή ε, ακόμη και πιο πέρα, αναλόγως με το για ποιο μέσο συγκοινωνία μιλάμε και ποια εναλλακτική ενέργεια. Βεβαίω ε, θα πρέπει να υπάρχει ο πυρηνά ε, πριν το 2030, θα πρέπει να υπάρχουν δηλαδή οι υποδομέ και πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι από τα δίκτυα TNT. Όμως λίγα πράγματα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Λάβουμε υπόψη το ότι μπορεί να πληρώσει το κάθε κράτο μέλο το τι είναι εφικτό, ε, για τα πάντα και για το υδρογόνο και για τα λοιπά καύσιμα. Θέλουμε βέβαια να έχουμε στο δυνατόν περισσότερο ανανεώσιμε πηγές και πράγματι έχουμε ε, αφενός την επιθυμία μα για αναθεώρηση, από την άλλη δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα στην εφαρμογή. Οπότε υπάρχουν ε, κονδύλια, υπάρχει το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, κάποιοι το έχουν ήδη κάνει, κάποια κράτη-μέλη σε κάποιους τομείς. Αλλά εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ λίγο και με αυτόν τον αριθμό δεν θα κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα το Κοινοβούλιο και να ασκήσει πίεση για να απομακρυνθούμε σιγά σιγά από τα όρεκτα καύσα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην ε, Κομισιόν, τον ε, κύριο Ντεπρέ. Αντικαθιστώ την κυρία Ντεπρέ βεβαίως που αποσιάζει με αρμόδιο στη Γενική Διεύθυνση μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τα μέλη της Επιτροπής. Συμφωνούμε πλήρως με όλα όσα ακούστηκαν. Γεγονός είναι πράγματι πως η βασική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να αυξηθεί ο συντονισμός ή η συνεργασία με τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή των εθνικών πλαισίων πολιτικής. Συμφωνούμε πλήρως ότι το επίπεδο συνοχής δεν είναι αυτό το οποίο θεωρούμε αναγκαίο, όμως, όπως είπαν σωστά κάποια κράτη-μέλη, κάποια, με συγχωρείτε, μέλη της Επιτροπής, πρέπει να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι δημόσιες υποδομές, φόρτισης έχουμε γύρω σε 130.000 σημεία φόρτισης ε, και 700.000 ε, οχήματα που μπαίνουν ε, στην μπρίζα. Βεβαίως δεν λαμβάνουμε υπόψη εδώ τις περιφερειακές διαφορές. Οπότε τώρα απευθυνόμαστε στην βιομηχανία να διαθέσει περισσότερα οχήματα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των καταναλωτών, να θέσουν ένα φιλόδοξο πλαίσιο τα κράτη-μέλη και να φροντίσουμε να πάμε προς μια διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αυτών. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να ταξιδέψει κανείς με ένα ηλεκτρικό όχημα διασυνοριακά, να βρει υποδομή και να ξέρει ότι θα λειτουργεί. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια τα οποία έχουμε, εργαζόμαστε σκληρά για είναι μια δράση προτεραιότητα στον επόμενο προϋπολογισμό. Προσπαθούμε ακριβώς ε, να αναμίξουμε τα διάφορα έργα υποδομών ε, και τέλος νομίζω πως είναι σημαντικό να δούμε τις ανάγκες διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και της αγοράς στην ε, Ένωση γιατί πρέπει πραγματικά να είναι σαφές ε, για τους καταναλωτές ότι είναι απλό να διασχίζει κανείς ε, τα σύνορα με ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα και θα πρέπει ακριβώς να έχουμε μια τεχνολογική ουδετερότητα και το φυσικό αέριο είναι μια καθαρή εναλλακτική για τις μεγάλες αποστάσεις και τέλος ε, ξεκινάμε με μια αξιολόγηση της οδηγίας αυτής. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εκθέσεις που πρέπει να μας στείλουν τα κράτη-μέλη. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τις ανάγκες αναθεώρησης της οδηγίας για να αυξηθεί και η αποτελεσματικότητά της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Τέλος, δίνω τον λόγο στον εισηγη... στην εισηγήτρα για δύο λόγια. Για δύο. Ευχαριστώ, ε, συνάδελφοι, για τα ε, σχόλιά σας. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι επί της ουσίας συμφωνούμε μεταξύ μας. Ελπίζω να υποβάλλετε κάποιες τροπολογίες έτσι ώστε η τροπολογία μας, η, συγγνώμη, η ε, γνωμοδότησή μας να καταστεί ε, ακόμα πιο αποτελεσματική. Και αν η Επιτροπή συμφωνεί μαζί μας, ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι σε αυτό το τομέα. Ε, τώρα υπάρχει μια προθεσμία για την επόμενη ε, Τρίτη για την υποβολή των τροπολογιών σας. Ελπίζω λοιπόν να τις υποβάλλετε έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε μια πολύ καλή ποιότητα γνωμοδότηση. Και βέβαια ελπίζουμε ότι αυτά τα ζητήματα που θα θέσουμε θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, 12 Ιουνίου ε, προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών. Ψηφίζουμε εδώ στην Επιτροπή μας στις 10 Ιουλίου, ενώ η ψηφοφορία στην Επιτροπή Τραν θα είναι στις 24 Σεπτεμβρίου. Ε, και σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής σας ε, διάταξης που είναι η ποιότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, αναδιατύπωση αυτής της ε, οδηγίας και βέβαια καθώς έχουμε υπερβεί λίγο το, το χρόνο που είχαμε προβλέψει θα προσπαθήσω να είμαι πολύ αυστηρός σε ό,τι αφορά το χρόνο αγόρευσης. Άρα λοιπόν θα δώσω το λόγο ε, στο για 5 λεπτά για να κάνει μια αρχική παρουσίαση. Μετά θα δώσω 3 λεπτά στους κοιόδης εισηγητές και 2 λεπτά στους υπολείπους συναδέλφους. Και βέβαια στο τέλος 5 ε, λεπτά και στην Επιτροπή καθώς και κάποιο χρόνο για να σχολιάσει καταληκτικά. Προφανώς θα ήθελα να υπάρξει περισσότερος ε, χρόνος ε, ε, για να συνεχίσουμε, αλλά θα πρέπει να διακόψουμε στις 12.30 ακριβώς. Οπότε δίνω το λόγο στον εισηγητό κύριο Νταντέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η πρόταση τη οδηγίας έχει στόχο να διορθώσει την πρώτη διόρθωση που έλαβε χώρα το 98 για το πόσιμο είδωρ που χρονομολογείται από το 1980 αρχική. Στην πρότασή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει βασικά να τροποποιήσει τη λίστα των παραμέτρων του προσήμου ύδατος. Προτείνει να γενικευθεί μία προσέγγιση βάσει του κινδύνου όσον αφορά την παραγωγή και διανομή του ύδατος. Συμπεριλαμβάνει αυτά που είχαν αναφερθεί από την πρωτοβουλία πολιτών, ενίσχυση της διαφάνειας δηλαδή και πρόσβαση των καταναλωτών σε πληροφορίες όσον αφορά το είδωρ που καταναλώνει και ξεκινά μια ευαίσθητη συζήτηση όσον αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό. Εν γέννη, πιστεύω ότι οι βελτιώσει και η προσέγγιση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι σωστή κατεύθυνση. Ευθυγραμμίζονται οι παράμετροι με την ποιότητα, της με τι επιστημονικέ έρευνε και δημιουργείται πιο στέρεο πολιτικό πλαίσιο για την προστασία των πηγών και ε, τη υγεία των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, σημείωσα και διάφορε ε, δυναμίε. Το κείμενο θεωρώ ότι λείπει, ε, λείπουν κάποιες πρακτικές πτυχές από την έκθεση και κάποιες επιτόπιες ε, πραγματικότητες όσον αφορά την εσωτερική διανομή του νερού, την υποχρέωση δειγματοληψίας παραδείγματος χάρη. Ε, πιστεύω ότι μια μελέτη που υποεκτιμά τον οικονομικό και χρηματοστατικό αντίκτυπο για τους παρόχους ύδατος και τελικά για τον καταναλωτή και καλό θα ήταν σίγουρα να το συζητήσουμε αυτό το σημείο. Η προσφυγή στην αρχή της πρόληψης θεωρώ ότι είναι κάπως επικριτέα όσον αφορά τις, αναδιόμε, τις ουσίες στην, στον ποιοτικό έλεγχο. Υπάρχει μια μίξη που χρειάζεται ξεκαθάρισμα στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι η διάθεση της οδηγίας με τις άλλες ε, νομοθεσίες Ευρωπαϊκής Ενώσης και στην οδηγία πλαίσιο για το είδωρο, αλλά όχι μόνο αυτό, ε, και όλα που σχετίζονται με τη χρήση του νερού στην επεξεργασία τροφίμων, όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν. Για αυτό το λόγο λοιπόν σας πρότεινα και κάποιες τροπολογίες που έχουν σαν στόχο ε, να τονιστούν τα διάφορα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού σύμφωνα με τις επιταγές του ΠΟΗ, Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν ποιες είναι οι διάφορες ευθύνες σε σχέση με το κείμενο τα κράτη-μέλη που έχουν ευθύνε να συμμορφωθούν με τι προδιαγραφέ για την ποιότητα του νερού, ε, θα πρέπει να βλέπουμε κατά πόσο αν ξεπερνιούνται κάποιε παράμετροι, δημιουργούνται επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, αν έχουν άμεση, άμεσο αντίκτυπο για την ανθρώπινη υγεία μέσω, αν ξεπεράσουμε κάποιε παραμέτρου και αν ξεπεράσουμε κάποιε άλλε παραμέτρου σε συνδυασμό με κάποια άλλα στοιχεία επηρεάσουν την υγεία. Αν χρειάζεται μια προσέγγιση εφοροποιημένη. Το σύστημα τη παρέκκλησης θα πρέπει να παραμείνει με προσαρμογέ στο παρόν πλαίσιο και ε, να οδηγεί σε πιο ταχεία συμμόρφωση των κρατών μελών. Αυτά όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα. Όσον αφορά τη γενίκευση της ε, προσέγγιση που βασίζεται στο ρίσκο, θα πρέπει να βασιστούμε στην αρχή ότι οι φορείς του ύδατος γνωρίζουν τα σωστά πλαίσια. Θα πρέπει να τηρήσουμε τα διάφορα χρονοδιάγραμμα που έχουν τεθεί για να μην πολλαπλασιαστεί η δειγματοληψία και να μειώσουμε το κόστος. Όμως παρόλα αυτά προτείνω να μην προχωρήσουμε πολύ μακριά όσον αφορά τους κινδύνους εντός των κατοικιών όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλα αυτά υπάρχουν κινδύνοι ε, που έχουν διαπιστωθεί στο χώρο που υποδέχεται εύθραυστο τμήμα του πληθυσμού όπως ε, διάφορες οικίες με υπερήλικες, ε, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και κέντρα συνεδριάσεων που δεν χρησιμοποιούν τακτικά, ε, δεν χρησιμοποιούνται τακτικά όπως είναι κέντρα συνεδρίων αλλά φιλοξενούν πολύ κόσμο. Αυτά χρειάζονται περισσότερη παρακολούθηση αλλά δεν πρέπει να παρακολουθούμε τι γίνεται σε κάθε κατοικία όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιούνται, πιστεύω ότι οι πρώτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στοχεύει σε μια τυποποίηση τύπου ε, ειδών για την κατασκευή, για την οικοδόμηση σπιτιών, Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν διαφορετική προσέγγιση. Έχουν κάνει κάποια κράτη-μέλη πρόταση στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να δούμε την πρόταση με ενδιαφέρον. Όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτικό νερό, χρειάζεται υψηλή ποιότητα για όλους, ε, με ε, χαμηλό κόστος και αυτό το θέμα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συνετής προσέγγισης, να μην φτάσουμε σε ακραίες λύσεις που θα διηγούσε σε μέτρα που δεν μπορούν να εφαρμοστούν όσον αφορά τις, ε, τη διαφάνεια τη πληροφορία στην ποιότητα του νερού. Πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των πληροφοριών που είναι γενικέ, που πρέπει να προσβάσουμε στο διαδίκτυο μονίμω και ενημέρωσης πιο διδακτικού περιεχομένου που μπορεί να βρει κανείς ε, στο λογαριασμό του νερού. Τώρα θέλω να ακούσω ότι έχουν να πούν οι σκιώδεις και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτος σκιώδης εισηγητής, ο κ. Φραν. Τρία λεπτά δεν είναι πολλά. Ε, είναι σημαντική οδηγία, καλύπτει πολλά ζητήματα, δεν μπορώ να καλύψω όλα τα σημεία που θα ήθελα. Εκ μέρους ομάδας μου θα ξεκινήσω με σημαντικότατο θέμα. Πολλοί από εμά θεωρούμε σαν δεδομένο ότι όταν ανοίξουμε τη βρύση, το νερό που βγαίνει από τη βρύση είναι πολύ συχνά καθαρό και ασφαλές. Και βεβαίως αυτό δεν ισχύει για όλους και δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να καθοδηγήσει την οδηγία και την προσέγγιση μας όσον αφορά αυτήν είναι ότι το 2018 στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε πολίτη παντού θα πρέπει να ασκεί το δικαίωμά του σε ασφαλές, φθηνό, καθαρό, πόσιμο νερό. Να πω ευθύ εξ αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την υποστήριξή μα για την ανανέωση αυτή τη οδηγία, ούτω ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα σημαντικά θέματα που αφορούν το δικαίωμα των πολιτών στο νερό, κάτι που έθεσε η πρωτοβουλία των πολιτών. Είναι κάτι που δεν πρέπει να λησμονούμε. Βέβαια εξυπακούεται, αλλά θα το πω, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι η ομάδα μας ε, θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποστηρίξει αδίποτε πρόταση της σχετικά με την οδηγία η οποία θα μπορούσε να ειδωθεί σαν μια αποδυνάμωση της δημόσιας υγείας και της προσέγγισης που ακολουθούμε για τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι βασικό σημείο όσον αφορά το, τις εργασίες μας επί της οδηγίας. Και θεωρώ ότι η καλύτερη πολιτική για τη δημόσια υγεία είναι η πολιτική που βεβαίως προστατεύει τη δημόσια υγεία αλλά δεν δημιουργεί ανησυχίες χωρί να χρειάζεται. Και χρειάζεται μια πολύ λεπτή ισορροπία. Και όταν θα εξετάζουμε τι λεπτομέρειε τη πρόταση, φαντάζομαι ότι θα πετύχουμε. Ε, θα, θα Πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να πετύχουμε τη λεπτή ισορροπία για να καταλήξουμε συμβαστικέ θέσει. Να πω εν συντομία κάποια παραδείγματα εν συντομία. Πρώτα απ' όλα, οι ενδοκρινικοί ε, διαταράκτε. Ανησυχεί ο κόσμο όλο και περισσότερο γι' αυτό. Έχουμε διάφορα στοιχεία που διαφαίνονται. Θα πρέπει να βρούμε μια συμβαστική λύση επ' αυτού που θα πρέπει να αναγνωρίσει την ύπαρξη λεπτή ισορροπία. Δεύτερο παράδειγμα. Το θέμα στη, κάποιων βρέθηκαν στην Ιταλία ε, και συνάδελφος Βάλλη το επεξεργάζεται. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί κατεύθυνση σωστή, ε, ο εισηγητής όμως ακολουθεί διαφορετική ε, κατεύθυνση. Αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε τις προσεγγίσεις για θέματα που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας. Δεν συμφωνούμε απαραίτητα με όλε τις προτάσει του εισηγητή. Σε αυτή τη φάση όμω θα πρέπει να παραδεχτώ ότι έχει καταβάλει Πολλέ προσπάθειε είναι διεξοδική εργασία του και προσβλέπουν στη συνεργασία μαζί του, ελέγχοντα τι προτάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, αναπτύσσοντας την ανταπόκριση του Κοινοβουλίου. Κλείνοντα, ξέρω ότι έχουμε χρονικά όρια, τα θέματα προσβασιμότητα ε, και τιμή του ύδατο είναι πολύ σημαντικά για μα. Στην ομάδα του SD θα υπάρξουν θέματα για τα οποία θα υποβάλουμε συγκεκριμένε ε, τροπολογίε για να ενισχύσουμε το κείμενο που έχουμε μπροστά μα. Διότι αν το νερό δεν είναι αρκετά φθηνό, τότε δεν είναι καν προσβάσιμο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόρμαν είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την ομάδα για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Η πρόσβαση στο πόσιμο νερό είναι πολύ σημαντική. Επηρεάζει την καθημερινή ζωή και την υγεία των πολιτών. Η ισχύουσα οδηγία δεν έχει αλλάξει εδώ και 20 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να την ξαναδούμε και θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, με τις ε, διαρροές. Είναι πολύ ψηλό το ποστό. 23% των ε, υδάτων χάνεται στους σωλήνες, κάπου στην διαδρομή. Και βεβαίως αυτό σχετίζεται και με την ε, υγιεινή. Όσο πιο πολύ χάνουν οι σωληνώσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα για μολυσμένο νερό. Ίσως ε, είναι πολύ φτηνό το πόσιμο νερό, γι' αυτό κανείς ε, δεν ενδιαφέρεται να λειτουργεί σωστά το σύστημα. Θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα όπου οι εταιρείε θα χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές ε, θα υπάρχουν ε, συγκρίσεις ε, και θα υπάρχει διαφάνεια. Και βεβαίως να υπολογίζουμε όχι μόνο την απώλεια του νερού αλλά και της ενέργειας. Δεν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα δίνει μεγάλα μερίσματα στους ε, μετόχους αλλά θα παρέχει καθαρό πόσιμο νερό και βλέπουμε πως το νερό ε, ρηπαίνεται εάν επιτρέπεται στις εταιρείες απλά να θάβουν δηλητήρια και σκουπίδια. Έτσι είναι δύσκολο το πράγμα. Τέλος ανησυχώ για την κοινωνική διάσταση που παρουσίασε η Κομισιόν. Η κοινωνική νομοθεσία είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Υπάρχει μια, μια ατύχης τάση δυστυχώς σε αυτό το μέτωπο και βλέπουμε ότι πρέπει να κάνουμε ε, τη δουλειά μόνοι μας ε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βακτηρίδια στο νερό. Ευχαριστώ κυρία Μελνέρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ και ε, αντιμετώπισε τις ελλείψεις ε, της πρότασης της Κομισιόν αλλά ευχαριστούμε και την Κομισιόν για τον πολύ επικοδομητικό διάλογο η οδηγία μου ύδατος είναι κάτι το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερος γιατί εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα αυτό ήδη από το επίπεδο του Δήμου που ήμουν πολιτικός για να μπορούμε να εγγυηθούμε καθαρό πόσιμο νερό. Στην Γερμανία έχουμε γύρω στους 6.000 παρόχους ε, δημοτικές επιχειρήσεις ε, υδάτων, κατά κανόνα δημοτικές. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει αυτή η προσέγγιση που θα βασίζεται στον κίνδυνο ε, αλλά να μπορεί να εφαρμόζεται και από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, ίδρυυσης. Και ακριβώς εδώ πέρα είναι το θέμα των παραμέτρων και της επίβλεψης που πρέπει να συζητήσουμε. Μια νέα καινοτομία της πρότασης της Κομισιόν είναι η ενημέρωση των καταναλωτών. Ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο προϊόν είναι οπωσδήποτε πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνεται ο καταναλωτής και είμαι σαφώς υπέρ. Όλες οι σχετικές ε, πληροφορίες για την ποιότητα του νερού πρέπει να είναι διαθέσιμες ε, με τρόπο απλό. Αλλά πρέπει νομίζω να συζητήσουμε ποιες είναι οι πληροφορίες που είναι όντως σημαντικές για τον καταναλωτή και ποιες βοηθάνε. Γιατί κάποια σημεία εδώ πέρα είναι σε λάθος. Ε, βάση. Επίσης θα ήθελα να στηρίξω τον ε, εισηγητή ε, για τον κατάλογο παρατηρήσεις για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες ή για τα μικροπλαστικά και επίσης το θέμα της σύνδεσης με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Δεν είναι σαφής εδώ πέρα η πρόταση της Κομισιόν σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, ξεκάθαρα πρέπει να προστατευτεί η επικουρικότητα. Είναι σημαντικό θέμα, όπως είπα, για τους Δήμους ε, η ίδρυυση, αλλά πρέπει να παραμείνει στα χέρια των Δήμων και να είναι, όπως είπαμε, το νερό πρόσιτο. Και χαίρομαι για την ε, συνεργασία. Είναι σημαντική οδηγία και πρέπει να γίνει προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ για τους πράσινους. Θα παρουσιάσω εγώ την θέση μας να ευχαριστήσω Κομισιόν και εισηγητή για την εξαιρετική τους δουλειά. Θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόταση της ε, Κομισιόν και συμφωνώ με πολλά από τα ζητήματα που ανέφεραν στην πρόταση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει ανανεωμένη λίστα χημικών ε, παραμέτρων. Επίσης είναι σημαντικό να δούμε το θέμα της μεγαλύτερης διαφάνειας και πρόσβασης ε, των καταναλωτών στις ε, πληροφορίες. Και βεβαίως συμφωνώ με τον εισηγητή εκεί όπου στην επεξηγηματική του έκθεση λέει ότι οι παράμετροι του παραρτήματος ένα είναι ε, ο θεμέλιος λήθος αυτής της οδηγίας. Από την άλλη, όταν ε, μπαίνουμε στις λεπτομέρειες, ε, πολύ απλά καταργεί κάποιες παραμέτρους ο εισηγητής, αυξάνει τα επίπεδα για κάποιες άλλες και υπάρχει δυνατότητα τα κράτη-μέλη να αποκλίνουν. Και από... και υπάρχει και μείωση των απαιτήσεων παρακολούθησης. Ε, προφανώς ε, δεν με ικανοποιούν ιδιαιτέρως αυτά. Παραδείγματο χάρη η ενδοκρινική διαταράκτηση είναι σημαντικό πρόβλημα και για το θαλάσσιο περιβάλλον και πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να τα δούμε αυτά τα ζητήματα όχι μόνο εδώ στην οδηγία αν δεν τα βάλουμε στον κατάλογο δεν θα γίνει και τίποτα σε σχέση με την οδηγία. Σε σχέση με τις ε, φθοριούχέ ε, ουσίες είναι περίπλοκο το ζήτημα γιατί η βιομηχανία ακριβώς ε, ασχολείται με την αλλαγή της μοριακής δομής αυτών των ουσιών και αντικαθιστούν τις ουσίες αυτές με πολύ παρόμοια μόρια και εάν επικεντρωθούμε μόνο στις ήδη απαγορευμένες ανοίγει η δυνατότητα για τη βιομηχανία να εισαγάγει νέα μόρια τα οποία δεν καλύπτονται τώρα για τις ενώσεις του χλωρίου και τον μόλιβδο δεν θεωρώ ότι οι παρεκκλήσεις που προτάθηκαν από την Κομισιόν δηλαδή να έχουν τα κράτη-μέλη την ευκαιρία να ε, εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της αρχικής οδηγίας ε, προετών ε, χρειάζονται και συμφωνώ ότι η διαφάνεια είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα η καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες ή διαφάνεια μας οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η οδηγία που συζητούμε σήμερα για το είδωρ που χορηγείται στον καταναλωτή ήταν ε, βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα ύδατα και συνάβαλε κατά πολύ για την ασφάλεια του πόσου νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλό να επικαιροποιηθεί τώρα και να κανονίσουμε ποιε είναι οι τιμέ αναφορά κάποιων χημικών και βιολογικών παραμέτρων. Λοιπόν, ευπρόσδεκτη η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επίτροπή ε, για να διατύπωση οδηγίας. Πιστεύω ότι κάποιε πτυχέ, κυρίω στο επιστημονικό τμήμα τη ε, προτάσεω, αντικατοπτρίζουν μια, συν, μια προσέγγιση ε, με προσοχή για να δώσει ένα ενισχυμένο καθεστώς ασφαλεία για του πολίτε βάσει τη αρχή τη πρόληψη και περνάει ακόμα και τα πλαίσια που προτείνει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Λοιπόν, το Ευρωκοινοβούλιο ε, πρέπει να είναι ικανοποιημένο από αυτή την προσπάθεια. Το αίτημα να αξιολογηθεί η παρουσία μικροπλαστικών ουσιών ε, και διαφόρων ενδοκρινικών διαταρακτών και σορευτική παρακολούθηση για διάφορες θωριούχες ουσίες. Τα φάσο όπως αποκαλούνται θα πρέπει λοιπόν να ε, υπάρχει προστασία όσον αφορά αυτές τις ουσίες που δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το περιβάλλον. Και παρουσιάζονται τα συμπτώματα βία κάμια φορά. Ε, όπως είδαμε και στην μεμόλυνση στην περιοχή του Βένετου στην Ιταλία. Λοιπόν, θα πρέπει να συνεργαστούμε επικοδομητικά για να βελτιώσουμε κάποιες στοιχές, όλος ιδιαίτερος οι διαταγέ όσον αφορά την προσέγγιση βαστού του κινδύνου και την αξιολόγηση του κινδύνου, πρέπει να καθορίσουμε καλύτερα τον ρόλο και την ευθύνη των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων. Πιστεύω ότι καλό περιθώριο βελτιώσεως υπάρχει στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το, την πρωτοβουλία των πολιτών για το δικαίωμα στο ίδρυμα, άρθρο 13 της πρότασης. Προσωπικά σαν Ιταλίδα πολίτης που το 2011 ψήφισε το δημοψήφισμα με πάνω από 27 εκατομμύρια Ιταλούς πολίτες υπέρ του δημοψηφίσματος για το δημόσιο είδωρ, δεν μπορώ παρά να δώσω μεγάλη σημασία στη δημόσια διαχείριση της υδροδότησης για να υπάρχει καθολική ε, πρόσβαση στο είδωρ που πηγαίνει μαζί με άλλα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει να υπάρχει ιδιωτικοποίηση. Απέτυχε ιδιωτικοποίηση της υδροδότησης στην Ιταλία αλλά και αλλού. Θα πρέπει να υπάρχει είδωρ προσβάσιμο σε όλους ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του καθενός. Θα πρέπει με την πρόταση που έχουμε και συζητάμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε σοβαρή ανάλυση όσον αφορά την απώλεια νερού κακή διαχείριση που οφείλεται και από την, ε, που επιδεινώνεται και από την αλλαγή του κλίματος. και υπάρχει απώλεια σε κάποιες περιοχές της χώρας μέχρι 60% του νερού από το δίκτυο χάνεται από απώλειες. Η κυρία Μπόιλαν είναι η επόμενη συνσηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, και ε, ζητώ συγγνώμη για την ε, καθυστέρησή μου εδώ, αλλά δεν είχα βέβαια τη δυνατότητα να περιορισκόμαι σε δύο ε, συνεδρία ταυτόχρονα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστώ τον ε, εισηγητή και τους, ε, τον εισηγητή και τους και εισηγητές για την τοποθετήσεις του εδώ. νομίζω πως είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε πως η οδηγία για το πόσιμο νερό ε, οδήγησε με κατάσταση όπου έχουμε σχετικά ασφαλέ νερό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο βέβαια θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Ε, Πάντω, ε, χαιρετίζω την εισαγωγή, την συμπερίληψη του άρθρου 13 στην πρόταση τη οδηγία, καθώ η σχετική πρωτοβουλία ήταν η μοναδική και έλαβε όχι μόνο ένα εκατομμύριο υπογραφών που είναι το απόλυτο ελάχιστο όριο, αλλά 1,9 εκατομμύρια. Οπότε γνωρίζω πως η Επιτροπή απάντησε κάτι πρώτα της αντίδραση ότι θα έκανε κάποιε προτάσει για να απαντήσει σε αυτήν την πρωτοβουλία ε, πολιτών. Ωστόσο, ε, το σύστημα του ΙΣΑΕ δεν αντιμετωπίζεται πλήρω με την πρόταση αυτή τη Επιτροπή. Οπότε, αποτελεί μια μερική μόνο απάντηση σε αυτήν την πρωτοβουλία που έγινε. Ε, η εν λόγω πρωτοβουλία αναφερόταν στα ζητήματα ιδιωτικοποίηση των σχετικών υποδομών, αλλά και στα ζητήματα αποχέτευση και ίδρυυση στο πλαίσιο τη του κανονιστικού πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καλό είναι το ότι γίνεται ε, ε, λόγο για την προσβασιμότητα στο πόσιμο νερό, ειδικότερα από ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού. Αλλά είναι από την άλλη πλευρά αδύνατο το να αναφέρεται κανείς σε ζητήματα προσβασιμότητας αν ε, δεν αναφερθεί ταυτόχρονα και σε ζητήματα ε, προσιτών τιμών. Δηλαδή αυτές οι δύο πτυχές πηγαίνουν μαζί και δεν είναι δυνατόν να αποσυνδεθούν η μία από την ε, άλλη. Γνωρίζουμε ε, πως ε, ε, ο Παγκόσμιος Οργάνωση Υγείας λέει πως το, κατά το μέγιστο 3% του προπολογισμού ενός νοικοκυριού θα πρέπει να δαπανάτε για το ε, <clears throat> πόσιμο νερό. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα ζητήματα ένες ό,τι αφορά το νερό τα οποία παραμένουν. Ε, οπότε ε, χαιρετίζουμε την αντίδραση από την πλευρά της ε, Επιτροπής σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών και βέβαια το αρχικό ψήφισμα από την πλευρά του Κοινοβουλίου που υποστήριξε τη σχετική πρωτοβουλία. Άρα λοιπόν η δική μου πρόταση και οι μου τροπολογίες αφορούν στην ενίσχυση του άρθρου 13 της πρότασης της Επιτροπής, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ πως είναι σημαντικό να επιχειρηματολογήσουμε και νομικώς ως προς το γιατί το άρθρο 1 της οδηγίας θα πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω. Γιατί ε, εάν με αυτόν τον τρόπο ανταποκριθεί η Επιτροπή ε, στην πρωτοβουλία των πολιτών, τότε και τα όσα προβλέπει ε, θα πρέπει να και αυτά με τη σειρά τους να ανταποκρίνονται. Και έτσι όπως είναι διατυπωμένη αυτή η οδηγία αυτή τη στιγμή δεν αναφέρεται παρκώς στα ζητήματα πρόσβασιμότητας. Επίσης χαιρετίζω αυτό που ε, αναφέρει η Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες πρόσβασης ε, στο πόσιμο νερό, αλλά με προβληματίζουν λίγο υποχρεώσεις ενημέρωσης ε, που προβλέπει. Για παράδειγμα, αυτές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 14 πηγαίνουν λίγο πέρα από το όσα καλύπτει το πεδίο εφαρμογή, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και κάποιο περαιτέρω άχθο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι τεχνικέ πτυχέ, θα προσπαθήσω. θα υποβάλω τροπολογίε σε, σε ό,τι αφορά ε, την, ε, τις προτάσεις για την ανθεώρηση του συστημάτων σε ό,τι αφορά τις, ε, το, ειδικότερα το ζήτημα των συγχρονότητων και από εκεί και μετά θα συνεχίσω να υποστηρίζω την προσέγγιση που έχει οθετήσει η Παγκόσμια Οργάνωση Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ να τηρείτε όλοι τις προθεσμίες σας γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Η κυρία Κοντέν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νταντέν για την έκθεσή του και τι διάφορε συστάσει ε, που μα υποβάλλει σήμερα. Καταρχά, να υπενθυμίσω ότι τα κράτη-μέλη και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι επιφορτισμένε για την πρόσβαση στο πόσιμο είδωρ. Αυτό είναι σχετικό και αποδίδει, λαμβάνει υπόψη τι ιδιαιτερότητε κάθε περιοχή και νομίζει ότι δεν πρέπει να διτηράξουμε την ισορροπία που σεβόταν ε, ε, η οδηγία του 1998. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει μια αναθεώρηση χωρίς να κάνει πραγματικές αλλαγές επί της ουσίας μέσω διατάξεων που θα οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους ε, για τον καταναλωτή. Επίσης, βασίζομαι στα κάτι μέλη και στο Συμβούλιο που θα εγγυηθούν την αρχή, το σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας στην συζήτηση φορά αφορά την αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας. Σχετικά με αυτό υποστηρίζω τις προτάσεις του εισηγητού για να αποφύγουμε την αύξηση της τιμής για τον καταναλωτή. Η βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πολλαπλασιάσει τα σημεία ελέγχου είναι κάτι κατανόητο. Εννοώ και οι συνθήκες για το πόσιμο χαρακτήρα της, ε, του ύδατος στην Ευρώπη ε, είναι κάτι που καλύπτεται και οι κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί μεγαλύτεροι. Δεν πεθαίνουν από χολέρα Ευρωπαίοι λόγω του νερού που καταναλώνουν. Και αυτό είναι υπέρ των φορέων υδροδότησης που εδώ και 40 χρόνια επεξεργάζονται το θέμα σε επιτόπιο επίπεδο ε, για, θα πρέπει να αλλάξουμε ίσως παράδειγμα και προσέγγιση και να μειώσουμε τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις πολυ... μικρές ουσίες όπως είναι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, τα μικροπλαστικά, διάφορες ουσίες κατάλοιπα φαρμάκων που σήμερα ε, δε, ε, μολύνουν ούτω ή πίν τον ορισμό του ποσίμου ύδατο. Χρειάζεται μια λύση για να αποφύγουμε αυτού του είδους ε, την ρήπανση. Η Λοζάνη δημιούργησε ένα σταθμό επεξεργασία υδάτων που ε, τα διάφορα κατάλοιπα φαρμάκων τα εξαλείφει. Λοιπόν, θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να θεσπίσουμε κάποιες διατάξεις για να ξανακαθορίσουμε την ποσιμότητα του ύδατος. Συμφωνώ με τον κύριο Νταντέν για το βασικό θέμα των ε, υλικών που έχω σε επαφή με το ίδρο και την πρόσβαση που έχει ο καταναλωτή σε πληροφορίε. Τέλο, όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβαση στο νερό, θα πρέπει να απαντήσουμε πλέον επακριβώ ε, όσον αφορά το τι σημαίνει αυτό. Θα αφήσουμε την πρωτοβουλία καλύτερα στα κράτη-μέλη. μη πέρα αυτού για την εφαρμογή και την ερμηνεία αυτού του δικαιώματο. Βέβαια, επ' αυτού δεν υπάρχει δωρεάν παροχή. Πάντα κάποιο ε, πληρώνει γι' αυτό και κυρίω ο φορολογούμενο. Ίσως θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε το γεγονότος ότι αυτό το δικαίωμα πρόσβαση στο νερό για όλους σημαίνει ότι το νερό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε λογική τιμή ε, και που θα υπάρχει ένα νότατο όριο της τιμής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στις ε, λοιπές παρεμβάσεις. Να σας θυμίσω ότι πραγματικά δεν έχουμε χρόνο. Δύο λεπτά το πολύ. Και να σας παρακαλέσω να είστε ακόμη πιο σύντομοι για να μπορέσει και ο ε, εισηγητής να απαντήσει. Ο κύριος Φλόρεντς, πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνω για τον χρόνο. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον εισηγητή, να έχει δίκιο και η Κομισιόν βεβαίως. Ε, προστίθενται νέες ουσίες η οδηγία είναι σχεδόν 20 ετών, οπότε καλά κάνουμε με δεδομένο του ότι έχουμε πλέον φάρμακα και μικροπλαστικά στο νερό και μια τέτοια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο είναι επίσης σωστή. Επίσης με ικανοποιεί το ότι η Κομισιόν δεν μπήκε σε ζητήματα πολιτικής και λέει να πίνουμε περισσότερο νερό από τη βρύση γιατί η συσκευασία και η μεταφορά τριών λίτρων νερού εμφιαλωμένου κοστίζει όσο 300.000 ε, λίτρα νερό της βρύσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω και να συνεχίσετε και βεβαίως να δούμε τα σημεία τα επίμαχα. Η εξέταση της ποιότητας ειδικά όσον αφορά τους ε, ιδιώτες ε, χρήστες ε, εκτός των δικτύων μου φαίνεται πολύ αυστηρή και τα υλικά τα οποία έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. Εδώ πέρα υπάρχει μια στρατηγική της Κομισιόν αλλά νομίζω ότι πρέπει να το αλλάξουμε για να μην τυποποιηθούν μόνο τα οικοδομικά υλικά αλλά όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. Βεβαίω, εντάξει, μπορούμε να οδηγηθούμε και στην υπερβολή. Ελπίζω λοιπόν να καταλήξουμε σε μία μέση προσέγγιση. Ευχαριστώ κύριο Ντεμέσμακερ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πω παρενθετικά ότι και το νερό που βγαίνει από τις βρύσες των Βρυξελών είναι εξαιρετικό οπότε μπορεί να αντικαταστήσει και τα πλαστικά μπουκάλια εδώ πέρα αλλά βεβαίως πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε για την ποιότητα. Συμφωνώ βεβαίως με τους αναγκαίους στόχους της αναθεωρησής αλλά τα σημεία κριτικής και αυτό που με ανησυχεί είναι κάποια τεχνικά ζητήματα που δεν έχουν ξεκαθαρίσει παραδείγματο χάρη πιθανή επικάλυψη μεταξύ αυτής της πρότασης και της υφιστάμενης ε, νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια στην νομοθεσία για να είναι ξεκάθαρο ποιοι κανόνες ισχύουν για ποιον κλάδο. Κατόπιν, βλέπω ότι η Κομισιόν στο παράρτημα 1 έχει άλλες τιμές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αλλά βλέπω πως το έχει επισημάνει και ο κύριος Νταντέν αυτό για τη δραστική αύξηση τώρα για την ε, παρακολούθηση και την ε, αφαίρεση διαφόρων ουσιών. Λοιπόν, ε, θεωρώ επίσης ότι ο κύριος Νταντέν πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση και οπωσδήποτε θα καταθέσουμε και κάποιες τροπολογίες με τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. εγώ να ευχαριστήσω τον συγκητή έξοχη δουλειά που έκανε. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την επιτροπή να βάλουμε το δάχτυλο από του σωστού τύπου των ύλων, να δούμε πιο ενθουσιαστικό, να εγγυηθούμε την ποιότητα του ποσίμου νερού στην Ευρώπη, που είναι απαραίτητη ανάγκη, χωρί να λάβουμε δυσανάλογα μέτρα. Διότι το κόστο θα επηρεάσει το λογαριασμό του καταναλωτή. Σχετικά με αυτό, λοιπόν, επιβάλλουμε καθημερινά ελέγχους ε, στο νερό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει νόημα, απόλυτο νόημα θεωρώ, να δοκιμάζουμε όσο χρειάζεται συχνά και συναρτήσει του κινδύνου του τόπου και συγκεκριμένη παραμέτρου θεωρώ ότι είναι πλέον δεδειγμένο. Πιστεύω ότι αυτή είναι η προσέγγιση που είναι προτιμότερη για τον εισηγητή. Άλλο θετικό στοιχείο, η επικαιροποίηση της επιστήμης ε, ε, για τις παραμέτρους αυτούς που έχουν, έχει ηλικία 20 ετών όπως ενδοκρινικοί διαταράχτες να ελέγχονται αν υπάρχουν και όχι μόνο αυτό και έχουμε σε μία ερώτηση που απευθύνω προς τον συγγετή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάλυση του κινδύνου που κάθε διανομέας νερού θα πρέπει να διεξαγάγει. Γιατί να βάζουμε διαφορετικές προθεσμίες εδώ ανάλογα με το μέγεθος του διανομέα. 3 ή έξι χρόνια. Χρειάζεται ισότητα μεταξύ των παρόχων και κυρίως η αρχή της ισότητας μεταξύ των καταναλωτών. Πρέπει όλοι να μπορούν να καταναλώνουν το πιο υγιές ε, νερό που μπορούν. Είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Η κυρία Σιαρπιέρικ, επόμενη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα σημαντικά αναφέρθηκαν ε, όσον αφορά και τις ε, εναρμονισμένες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό. Είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο και επίσης οι τερμολογίες γύρω από το σημείο 10 και βεβαίω ε, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή αντιμετώπιση των προσωρινών υπερβάσεων των ε, τιμών. Κατά λοιπά θα ήθελα να ζητήσω όπως συνήθως να γίνει σεβαστή η επικουρικότητα και να μην οδηγηθούμε βεβαίως σε μια υπερβολική νομοθέτηση πέρα από την νομική μας βάση. Και εδώ πέρα θα πρέπει να συμφωνήσω με την Γερμανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος όσον αφορά τις ουσίες PMT, οι οποίες, ε, τις οποίες αντιμετωπίσαμε επίσης και στο πλαίσιο της οδηγίας REACH. Ε, Αλλά θα θέσω και γραπτές ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γραμματικάκης. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι η Ήπειρός μας δεν αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου. Υπάρχουν όμως πολλά κρίσιμα ζητήματα που πριν είναι αργά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όπως για παράδειγμα προβλήματα υποδομών. Οι πολίτες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης, πρόσφατα στερήθηκαν για 10 περίπου μέρες το πόσιμο νερό. Ακόμα θέλω να αναφέρω ότι πολλές περιοχές της Ευρώπης, ιδιαίτερα τουριστικές, που ο πληθυσμός βέβαια πολλαπλασιάζεται κατά την τουριστική περίοδο, αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις πόσιμου νερού, με αποτέλεσμα οι πολίτες να στρέφονται στα εφιαλωμένα νερά με τα γνωστά αποτελέσματα που είπαν και άλλοι ομιλητές. Η κλιματική αλλαγή επίσης παίζει και εδώ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει δυστυχώς να είμαστε έτοιμοι για μια έγκαιρη προσαρμογή σε καταστάσεις εντονότερης ξηρασίας. Συγκεκριμένα επίσης κάποιες περιοχές δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών τους χαρακτηριστικών όπως είναι για παράδειγμα τα ελληνικά νησιά. Θα ήθελα όμως επίσης να θίξω και ένα θέμα που είμαστε πολύ ευαίσθητοι όπως φάνηκε και από τη μεγάλη πρωτοβουλία με τα δύο εκατομμύρια υπογραφές. Δεν υπάρχει κάποιος πιστικός, οικονομικός ή κοινωνικός λόγος για να υποστηρίξει κανείς την ιδιωτικοποίηση του νερού. Δυστυχώς όμως, να το τονίσω, στην περίπτωση του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής δηλαδή και με την έγκριση, λυπούμε να το πω, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι επιχειρήσεις ιδρεύσεως έχουν μπει στο λεγόμενο υπερταμείο, που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη τους. Σίγουρα, όπως είπαν και άλλοι ομιλητέ, θα ήταν πολύ καλύτερο να αφήσουμε τις τοπικές κοινωνίες να αποφασίσουν για την τύχη του νερού και του δικαιώματος του ανθρώπου. Thank you very much. And the last speaker is Mr. Haitama. Τελευταίος ο κύριος Χαϊταμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Είναι απαράδεκτο η Κομισιό να διαγράφει εδώ το άρθρο 10. Πρέπει να βασιστούν περισσότερο στο άρθρο 10 και να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό, να είναι χαμηλού κινδύνου και να υπάρχει μία εναρμόνιση. Πρέπει να εναρμονιστούμε και χαίρομαι που ο εισηγητής ακολουθεί αυτήν την γραμμή. Επίση το θέμα των παρεκκλήσεων για το άρθρο 9, παραδείγματο χάρη, δεν πρέπει να διαγραφεί, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν κάποιε παρεκκλήσει. Ομοίω και στο άρθρο 12 πρέπει να είναι σαφές αν υπάρχει μια προσωρινή υπέρβαση κάποιων παραμέτρων ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία. Μετά, πολλά ακούστηκαν ε, για την παρακολούθηση των διαφόρων παραμέτρων και την, προ... και την πληροφόρηση. Κοιτώντα την πρόταση της Κομισιόν, ναι, μπορούμε να παρακολουθούμε ε, και 365 μέρες το χρόνο, αλλά για ποιο λόγο. Ε, πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει. Χρειαζόμαστε ασφαλέστερο νερό, πρέπει να έχουμε λοιπόν μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου και θα, υπάρχει και, θα έχει και ξεκάθαρα εργαλεία διαχείρισης όχι επειδή μας αρέσει κάτι θεωρητικά να παρακολουθούμε διαφορετικές παραμέτρους επίσης η παροχή πληροφοριών ε, προς τις Βρυξέλλες ε, για ποιο λόγο ναι, έχει λόγο δεν υπάρχει λόγος να αυξάνεται η γραφειοκρατία για τις ε, εταιρείε ε, υδάτων αν δεν ε, αυξάνεται η ποιότητα του νερού. Λοιπόν, επειδή θα τελειώσει η ερμηνεία στο 12.30 ακριβώς, θα ήθελα να δώσω τον λόγο πρώτα στον εισηγητή και μετά στην Κομισιόν που θα μιλήσει αγγλικά. Ο κ. Νταντέν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους όσους παρενέβησαν. Πιστεύω ότι η συζήτηση συμπεριλαμβάνει τις θέσεις ε, που ήξερα από συνομιλίες με τους διαφόρους. Προσωπικά θα φροντίσω τόσο σώσο το κείμενο να παραμείνει επί του στόχου του. Κάποιες παρεμβάσεις προσπάθησαν να επανεισάγουν στο κείμενο πράγματα που δεν έχουν σχέση με αυτό το κείμενο. Μετά, επί επιστημονικής βάσης, μπορούμε να συζητήσουμε μεταξύ μας και να συμφωνήσουμε στο βαθμό του δυνατού. Ε, όταν συμφωνεί και επιστημονικό, επιστημονική κύκλοι συμφωνούν και με τα επιχειρήματά μας. Ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Μαργκά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα ε, τον εισηγητή, του και εισηγητέ και βεβαίω όλου σα που συμμετέχετε σε αυτέ τι εργασίε για την άριστη συνεργασία και διεξοδικό έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει ανοιχτή στη συνέχιση του επικοδομητικού διαλόγου και της μεθόδου εργασία που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Το δεύτερο που παρατηρώ από όλες τις παρεμβάσεις νομίζω σχεδόν ανεφεξαιρέσεων είναι ότι το γενικό πνεύμα της ε, προτάσεως και οι στόχοι που έχουμε προτείνει ε, είναι αποδεκτοί και στηρίζονται, αλλά βεβαίως ε, εδώ ακούγονται διάφορες απόψεις επαρκετών στοιχείων και θα ήθελα ίσω να μην κολλησιεργήσω, να μην καθυστερήσω, να διευκρινίσω δύο ζητήματα που ίσως μα βοηθήσουν σε μελλοντικέ συζητήσει, να επενδυμίσω του στόχου και μετά ε, να αναφερθώ σε κάποιε από τι αδυναμίες ε, που βλέπουμε στην έκθεση του συγητού και που τροφοδότησαν και κάποιε από, ε, από τα σχόλια των σκιωδών. Να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραμείνει πάρα πολύ επικοδομητική. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα που μέχρι τώρα μέσω της προτάσεως με σκληρή δουλειά μπορεί να εθετηθεί ε, σε αυτή τη θητεία και θα κάνουμε τα πάντα ό,τι μπορούμε για να το υποστηρίξουμε ε, και, στο, και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πάνω σε αυτό. Αυτό στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε είναι να παραμείνουμε πραγματικοί στους στόχους όπως είπε η Εδώ οι διερμηνεί πρέπει να σα πληροφορήσουν με τα λύπηση ότι συνεχίζεται η εργασιακή διαμάχη με τη δίκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι νέε συνθήκε εργασίας που αποτέλεσε αντικείμενο προειδοποίηση για απεργιακή κινητοποίηση. Η ποιότητα διερμηνία για του Ευρωβουλευτέ και του Ευρωπαίου πολίτε κινδυνεύει. Δυστυχώ, λόγω τη εργασιακή διαμάχη, η διερμηνία θα σταματήσει τώρα ακριβώ όπω προβλέπει το πρόγραμμα τη συνεδρίαση. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σα.